Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Με την δευτεριάτικη καθυστέρηση θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Κυρίσω την έναρξη της ε, συνεδρίας Επιτροπής μας. Η σε διάταξη. Με αίτημα τη ηγήτρια συντάκτηρα γνωμοδότη κυρία Κατεμπάχ, το σημείο 6 τη σε διάταξη, δηλαδή τη θάσευση ή αξιοποίηση τη ε, παγκοσμιοποίηση και οι εμπορικέ πτυχέ τη, ε, μεταφέρθηκε ε, για συζήτηση αύριο το πρωί, τρίτη πρωί δηλαδή, μετά το σημείο 11. Η ψηφοφορία το σημείο που αφορά τον εκτελεστικό κανονισμό για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα αναβάλλεται για μελλοντική συνεδρίαση της Επιτροπής. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις για την ημερήσια διάταξη και τις αλλαγές που σας πρότεινα, θα μπορούσαμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Επόμενο σημείο. Έχουμε διερμήνει από και προς 20 γλώσσες, με εξαίρεση τα τσεχικά, μαλτέζικα, σλοβακικά και γοεδελικά, κελτικά. Ενώ αύριο το απόγευμα που θα έχουμε τη συνάντηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια θα έχουμε διερμηνία από και προς 23 γλώσσες. Μόνο τα Ιρλανδικά δηλαδή θα έχουμε. Έγκριση των πρακτικών έγκριση πρακτικών των συνεδριάσεων τη 21ης και 22ης Φεβρουαρίου και 27ης Φεβρουαρίου. Όσοι αν δεν υποβληθούν παρατηρήσει μέχρι το πέρας της ε, συνεδρίαση, ε, θεωρούνται συγκεκριμένα τα πρακτικά. Περνάμε στο σημείο 4 που είναι το πρώτο ουσιαστικό ζήτημα της ημερήσιας διάταξης και θα ήθελα ευκαιρία, να καλωσορίσω θερμότατα στην Επιτροπή μας τον κύριο Ζωάου Φιγκερέντο, που είναι μέλος του πρώτου τμήματος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Καλώς ήρθατε κύριε Φιγκερέντο και εσείς και οι συνεργάτες σας. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας και θα ήθελα να τονίσω ότι αυτές οι ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι πολύ σημαντικές γιατί πραγματοποιούν μια ευρυθή ανάλυση ουσιαστική της κατάστασης και ε, συμβάλλουν στην ενίσχυση της συνεργασίας μας, γιατί αξιοποιούμε την τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη του ελεκτικού συνεδρίου και περιμένουμε με ενδιαφέρον τις στάσεις και προτάσεις γιατί εμείς έχουμε άμεση επαφή με τους γεωργούς και γι' αυτό με τα δικά σας φώτα παρακολουθούμε καλύτερα την εκτέλεση της κοινή γεωρικής πολιτικής. Ε, ο κύριος Φιγκερέντο και το επιτελείο του εκπώνησαν την ειδική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου με θέμα ένα πολύ σημαντικό θέμα για την κοινή γεωρική πολιτική, το καθεστώς της βασικής ενίσχυσης που αποτελεί και ένα από τα θεμελιώδη εργαλεία μέσα της κοινή γεωρικής πολιτικής. Πρόκειται για ένα καθεστώς, ένα μηχανισμό που στηρίζει άμεσα το γεωργικό εισόδημα και προσπαθεί να καλύψει αυτές τις ανισορροπίες που είναι αιτία πολλών προβλημάτων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και οι νεαροί αγρότες μεταξύ άλλων και ούτω καθεξής. Αυτές οι αιτήσεις δαπάνες της κοινή γεωρικής πολιτικής ε, από το καθεστώς βασικής ενίσχυσης είναι αρκετά σημαντικές. Και ε, πηγαίνουν στις συγκεκριμένες χώρες και στους συγκεκριμένους γεωργούς. αποτελώντας ε, σημαντικές και τακτικές οικονομικές ροές για τους αγρότες μας. Σε ό,τι αφορά τη συστηματοποίηση αυτού του καθεστώτος ε, βασικής ενίσχυσης, λαμβάνονται υπόψη και στην ε, μεταρρύθμιση της κοινή γεωρικής πολιτικής. Θέλουμε αυτές, αυτές οι βασικές ενισχύσεις να στηρίξουν το γεωρικό εισόδημα, σίγουρα, αλλά να μην ε, υπαγορεύουν συγκεκριμένες λύσεις ως προς ε, το μέσο και το προσανατολισμό, τα χαρακτηριστικά της παραγωγής που εξαρτάται από τις συνθήκες αγοράς περισσότερο. Περισσότερο το καθεστώς βασικής ενίσχυσης στηρίζει το γεωργικό εισόδημα. Φαντάζομαι όμως εσείς κύριε Φικερέντο θα μας τα πείτε πιο διεξοδικά κατά την παρουσίαση της έκθεσής σας. Σιγά σιγά γεμίζει και η αίθουσα. Έχουν έρθει στο μεταξύ όλοι οι συντονιστές από όλες τις πολιτικές ομάδες. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε κύριε Βραβουλευτέ, καλώς ήρθατε συνεργάτες, καλεσμένοι. Μπορούμε τώρα να δώσουμε το λόγο στον καλεσμένο μας, τον κύριο Ζωάν Φιγκερέντο, για να μας παρουσιάσει την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ε, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Για, το θερμό σας καλωσόρισμα και θέλω να πω ως μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η δική μα στάση και νοοτροπία είναι πάντα να είμαστε στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υποβολή των αποτελεσμάτων τη δουλειά μα. Με την ελπίδα ότι τα ευρήματα αυτά, ότι η δουλειά μας θα σας είναι χρήσιμη στο νομοθετικό σας έργο, στη χάραξη πολιτικής. Αυτή είναι η στάση και η νοοτροπία μας. Στη διάθεσή σας να προσφέρουμε όλη μας τη γνώση, τα ευρήματα, και τα απορίσματα της εργασίας μας. Κατόπιν της γενικής πρόσκλησής σας για υποβολή της ειδική έκθεσης για τα βασικά συστήματα πληρωμής για τους ε, γεωργούς, θέλω να παρουσιάσω τα κύρια συμπεράσματα. Πρόκειται για ένα μακροσκελές έγγραφο με πολύ λεπτομερείς πληροφορίες που μπορεί να είναι χρήσιμο για τη δουλειά σας. Κατά τη διάρκεια όμως της συνεδρίασης σκοπεύω να παρουσιάσω μόνο τα κύρια ευρήματα και συμπεράσματα. Έχω μία παρουσίαση σε PowerPoint για να καταστεί πιο σαφής η πληροφορία, το σύνολο των πληροφοριών που έχουμε ετοιμάσει. Τα συνολικά λοιπόν αποτελέσματα καταρχάς ε, του δημοσιονομικού ελέγχου είναι ότι το βασικό σύστημα πληρωμών, όπως εγκρίθηκε με τη μεταρρύθμιση του 2013, βασικό σύστημα λοιπόν πληρωμών για τους γεωργούς, ακολουθεί λειτουργικά ε, τον προγραμματισμό του, ωστόσο έχοντας υπαλληθεύσει με τη δουλειά μας και στα κράτη-μέλη και σε κάποιες υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με κάποια ερωτηματολόγια που απεστάλησαν στα κράτη-μέλη, διαπιστώνουμε ότι δεν συμβάλλει τόσο στην απλοποίηση, το ιστόχοποίηση και την σύγκληση των επιπέδων των ενισχύσεων. Αυτά λοιπόν είναι τα δύο αλληλοεξισορροπούμενα συμπεράσματα ότι το σύστημα το οποίο εγκρίνατε το 2013 ακολουθεί ε, το τον προγραμματισμό του, αλλά με περιορισμούς ως προς τα αποτελέσματα σε αυτούς τους τρεις τομείς, την απλοποίηση του στόχου, τη στόχοποίηση και την ε, σύγκληση των επιπέδων των ενισχύσεων και θα δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Σε σχέση με τους υπολογισμούς, για την ε, χορήγηση των ενισχύσεων βλέπουμε ότι καταβάλουν σημαντικές προσπάθειες οι υπηρεσίες πληρωμών. Διαπιστώνουμε ότι τα συστήματα ελέγχων στα κράτη-μέλη που επισκεφθήκαμε σε μεγάλο βαθμό περιορίζουν τον κίνδυνο ε, ανακριβών υπολογισμών και καταλογισμού ε, ενισχύσεων και ότι γενικά και σε επίπεδο ουσιαστικό δεν είχαμε σημαντικά σφάλματα στις ε, ενισχύσεις. Ωστόσο, ε, τα ποσά έχουν σε μερικές περιπτώσεις υπολογιστεί κατά τρόπο ανακριβή ή μόνο προσωρινό ή με βάση εκτιμήσεις. Και ορισμένες υπηρεσίες που επισκεφθήκαμε αντιμετώπισαν συγκεκριμένε δυσκολίες στους υπολογισμούς τους. Σε σχέση με τη γενική διαχείριση των πληρωμών και ξέρετε ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα κοινό μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρατών μελών. Βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει στα κράτη-μέλη κατευθύνσεις, οδηγίες και ελέγχους με καλά αποτελέσματα. Κάποιες πληροφορίες, ωστόσο, από την επιτήρηση βλέπουμε να απουσιάζουν. Ως προς δε τους φορείς πιστοποίησης, θεωρούμε ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να έχει ε, εκφράσει περισσότερες απαιτήσει στις υπηρεσίες αυτές των κρατών μελών. Ως προς την απλούστευση. Διαπιστώνουμε, όπως και εσείς φαντάζομαι θα έχετε αντιληφθεί, ότι η Διατάξει και κανόνε που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπουν πολλά ε, σημεία κατ' επιλογή ρυθμίσεων και εξαιρέσεων. Οι επιλογέ, πολλές επιλογές, ξέρετε, δεν διευκολύνουν την κατάσταση πάντοτε και δεν την απλοποιούν, γιατί οδηγούν σε διαφορετικέ λύσει τα κράτη-μέλη, οι οποίε δεν διευκολύνουν την απλοποίηση. Το δείχνουμε αυτό και στην έκθεσή μας, με παράδειγμα, στις γεωργικές περιοχές συγκεκριμένου κράτους μέλους που δείχνουν ένα πολύ περίπλοκο σχήμα. Κάποιες από αυτές τις επιλογές επιτρέπουν στους ορισμένους γεωργούς να εξασφαλίσουν επιπλέον κέρδους. Αυτό το επισημαίνουμε στην έκθεσή μας και πρόκειται για τα κύρια συμβράσματα που αφορούν τον τομέα της απλοποίησης. Ως προς την στόχευση, και βέβαια γνωρίζετε πως κύριος στόχος της μεταρρύθμισης του 2013 ήταν η καλύτερη στοχοποίηση ε, και εξυπηρέτηση των στόχων της πολιτικής μέσω των ενισχύσεων. Ω προ την εξυπηρέτηση λοιπόν των στόχων, διαπιστώνουμε και σας υπενθυμίζω μία νέα έννοια του ενεργού γεωργού που εισήχθη κατά τη μεταρρύθμιση του 2013. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποια θετικά αποτελέσματα. Εν γένει ωστόσο, σε σχέση με αυτή την έννοια του ενεργού γεωργού. Ωστόσο όμως, παρά τα καλά αποτελέσματα, ήταν δύσκολο να υλοποιηθούν και είχαν περιορισμένο αντίκτυπο. Όπως γνωρίζετε, από το, το νέο έτος, από το 2018, μπορούν τα κράτη-μέλη να περιορίσουν τα κριτήρια με, με βάση τα οποία ο ετών μπορεί να αποδείξει το καθεστώς ενεργού ε, αγρότη ή να διακόψουν, να κλείσουν τον κατάλογο. Ως προς τη στοχοποίηση και την εξυπηρέτηση των στόχων, έχει επεκτείνει τις κατηγορίες ε, για τη γη για τις οποίες μπορεί να καταβληθεί ενίσχυση και απαιτείται ελάχιστη γεωργική δραστηριότητα με βάση τη μεταρρύθμιση. Κάποια προχώρησαν περισσότερο στον περιορισμό του κινδύνου των κερδοσκοπικού χαρακτήρα ε, απαιτήσεων και αιτήσεων. Ωστόσο βλέπουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες στην υλοποίηση πάλι. στο θέμα της σύγκλησης των επιπέδων ενίσχυσης. Τα κύρια συμπεράσματά μας είναι τα εξή. Η μεταρρύθμιση του 2013 με τα επίπεδα ενίσχυση ανά εκτάριο καθιστά τις λύσει αυτές πιο ομοιόμορφες. Ωστόσο, σημειώνουμε ότι 11 από τα 18 κρατημάλη παρουσιάζουν ακόμη σημαντικέ ε, διαφορές, οι οποίες θα συνεχιστούν και μετά το 2019. Και εδώ σας δείχνω την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τα διαφορετικά μοντέλα σύγκλησης, ως προς τη σύγκληση μάλλον μεταξύ των κρατών μελών. Έτσι λοιπόν το σύστημα πληρωμών έχει περιορισμούς ως προς την αντιμετώπιση των προβλημάτων των εισοδηματικών των γεωργών και τίνει να ευνοεί τις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις. Επίσης, καθώς δεν υπάρχουν ε, στόχοι σαφείς, και τα επίπεδα είναι δύσκολο να οριστεί ε, η αποτελεσματικότητα και το πεδίο της ε, ενίσχυσης που προσφέρεται. Έτσι λοιπόν οι συστάσεις μας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνουν τα εξή. Πρέπει να αντιμετωπιστούν από πλευρά της Επιτροπής οι διάφορες αδυναμίες στα κύρια σημεία ελέγχου. Πρέπει η Επιτροπή να διορθώσει τις, ε, τα σημεία όπου οι αξίες έχουν σημαντική σημαντικό ποσοστό σφάλματο ή μπορούν να επηρεαστούν από εσφαλμένες πληροφορίες. Πρέπει επίσης να αναθεωρήσει τα συστήματα για την ε, ε, κοινοποίηση των πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών, να ενισχύσει την ε, κοινοποίηση κύριων πληροφοριών και να διευκρινίσει τους ρόλους που θα που θα επομίζεται είτε η Επιτροπή αφενός είτε οι αρμόδιες αρχές αφετέρου, οι τοπικές αρχές. Επίσης και τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει πριν από κάθε νέα πρόταση για το μελλοντικό σχεδιασμό της κοινή γεωργική πολιτικής να αναλύσει το ενδεχόμενο ενίσχυσης ε, εισοδηματικής για όλες τις ομάδες γεωργών και να ορίσει λειτουργικούς στόχους για οδήποτε μηχανισμό ενίσχυσης εισοδήματος, εξετάζοντας πώς μπορεί αυτός να σχεδιαστεί ώστε να ικανοποιήσει καλύτερα τους στόχους. Και επίσης θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε σχεδιαζόμενο και προτεινόμενο μέτρο να το συσχετίσει με λειτουργικούς στόχους και ε, κατώτατα όρια, βασικές γραμμές, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα σύγκριση με τις επιδόσεις και τον αντίκτυπο της ενίσχυσης. Αυτά κυρίες και κύριοι ήταν τα κύρια συμπεράσματά μας συμπεράσματα από το έργο του Μεσονομικού Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αυτά, ε, αυτές είναι οι συστάσεις που απευθύνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να λειτουργήσει καλύτερα στο μέλλον η κοινή γεωργική πολιτική. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Φιγκερέντο. Περνάμε τώρα στην Ομίγυρη. Πρώτο ο κύριος Αλμπερντές, ο συντονιστής του ΕΛΚ. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ τον Ελληνικό Συνέδριο για την έκθεσή του. Αντίθετα από το, η αντίστοιχη έκθεση για την οικολογικοποίηση, πρέπει να πω ότι εδώ βλέπω πράγματα πολύ λογικά, ε, γιατί στην έκθεση για την ε, οικολογικοποίηση βλέπουμε ότι χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση και έχω αποστείλει και επιστολή στον ε, πρόεδρο Λένε του ελεγκτικού συνεδρίου για την οποία νομίζω πρέπει να συζητήσουμε περισσότερο. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω το ελεγκτικό συνεδρίο να υπολογίζει τις γεωργικές δαπάνες ως ένα ποσοστό και να τις καταγράφει ως ένα ποσοστό των γενικών δαπανών του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού για να βλέπουμε την αναλογία στις εκθέσεις αυτές. Αυτό είναι το ένα που θα ήθελα να ζητήσω. Επίσης, δεν βλέπω παραπομπή στην πενταετία για τη μόνιμη οικολογικοποίηση, που θεωρώ ανοησία και πιστεύω ότι στην προσεχή μεταρρύθμιση και στο μέσο ε, προσεχές χρονικό διάστημα θα πρέπει να βρούμε άλλες λύσεις που θα είναι επαφέλεις για το περιβάλλον αλλά και για τους γεωργούς. Στην έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου, από ό,τι βλέπω και από την ε, συνοπτική παρουσίαση, τα, ε, υπάρχουν μόνο μονοκράτη κράτη-μέλη τα οποία προχωρούν σε ενιαία ενίσχυση το 19 και άλλο ένα το 20 η Γερμανία το 2019 θα έχει ενιαία ενίσχυση σε όλες τις εκτάσεις ανεξαρτήτως ε, ομόσπονδου κρατηδίου ή ποιότητα ε, του εδάφους. Και καλό βεβαίω όλα τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν την ίδια πορεία. Γιατί? Γιατί εάν δεν είχαμε αυτές τις πληρωμές με την κρίση στο γάλα, πολλές από τις ε, γαλακτοπαραγωγικές μονάδες θα είχε χρειαστεί να κλείσουν. Η Γερμανία χρειάστηκε 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ να τα ρίξει στο πρασίνισμα, στην οικολογικοποίηση. Εδώ λοιπόν χάσαμε ένα σημαντικό κομμάτι ενίσχυσης για, την, ε, για το γάλα. Και πιστεύω ότι και η κυρία Μίλλερ που ε, ασχολείται και αυτή με την ε, παραγωγή του γάλακτος θα έχει να πει αντίστοιχα παρατηρήσεις. Επίσης, για ε, τις αθμιστικές ε, πληρωμές ε, μπορούν να δώσουν κάποιες λύσεις. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό που λέτε και ενδιαφέρον. Θέλω επίσης να σημειώσω, άλλωστε το έχω επισημάνει και άλλες φορές, ότι το 1961 ε, πήρα δίπλωμα ε, οδήγησης για τρακτέρ γεωργικό, 14 ετών. Μου κόστησε ελάχιστα, 55,27 γερμανικά μάρκα τότε. Αυτό δεν είναι πλέον δυνατό. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει αυτή η δυνατότητα και πρέπει να είμαστε σε θέση, εάν πουλάμε κάτι σε τιμές του 1961, να έχουμε και την αντίστοιχη ενίσχυση σε τιμές του 1961. Και γι' αυτό θα ήθελα να δω εάν έχετε τις αναλογίες στα ποσά. Είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει στο μέλλον. Και νομίζω θα πρέπει να κοιτάξουμε μια πιο ισοδική κατανομή στα ποσά. Ευχαριστώ πολύ για την έκθεση. Είναι ενδιαφέρουσα. Είναι μια πολύ καλή βάση για περαιτέρω δουλειά. Ευχαριστώ κύριο Σαντρία. Προς το παρόν δεν περιορίζω το χρόνο αγόρευσης, αλλά δείξτε κάποια αυτοσυγκράτηση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο και τον εκπρόσωπό του για την υψηλή ποιότητα ε, έκθεση και το έργο του. Πράγματι δεν συμφωνώ με τον συνάδελφο Ντέ 100% για αυτά, σε αυτά που είπε για την οικολογικοποίηση, αλλά πράγματι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε. Είχαμε μια ε, έκθεση αυτή. Και επίσης γενικότερα για την αγροτική ανάπτυξη έρχονται οι εκθέσεις η μία μετά την άλλη. Ίσως θα έπρεπε να έχουμε μία συζήτηση στην οποία να τη συνθέσουμε, να δούμε τη συνολική εικόνα. Όλα δηλαδή, όλες δηλαδή τις πτυχές της κοινή αγροτικής ε, πολιτικής, έτσι ώστε να μην βλέπουμε αποσπασματικά την κάθε έκθεση, αλλά συνολικά το, το πρόβλημα. Ε, και πιστεύω ότι αυτό θα είχε πράγματι μια σημαντική προστιθέμενη αξία για το έργο της Επιτροπής μας. Φαίνεται λοιπόν ότι πρέπει, μια και θα ετοιμάσουμε την επόμενη ΚΑΠ, να δούμε τι ενισχύσει όχι μόνο από πλευρά ε, τη επίπτωση που έχουν στο αγροτικό ε, εισόδημα, αλλά και τι άλλε πτυχέ του. Δηλαδή, βεβαίω ότι πρέπει να φροντίσουμε τη διατροπιφική ασφάλεια, βεβαίω πρέπει να δούμε τι επιπτώσει τη ε, γεωργικής γεωργική παραγωγή στο περιβάλλον, Και τελικά όλα αυτά συντίθεται και μας ε, δίνουν το βασικό ερώτημα που είναι ποιο μοντέλο γεωργίας θέλουμε. Δεν μπορούμε να θέσουμε ε, στόχους όπως ζητάτε, όπως χρειάζεται, εάν δεν έχουμε απαντήσει πρώτα στο βασικό ερώτημα τι είδους γεωργία θέλουμε. Και σήμερα λοιπόν, 23 Απριλίου, έχουμε τις ε, συστάσεις σας ενώ στις 29 περιμένουμε την πρόταση της Επιτροπής, η 2 Μαΐου, και αναρωτιέμαι πώς μπορούμε με αυτό το τόσο πιασμένο χρονοδιάγραμμα να συνεισφέρουμε σε, μια, σε έναν εξυγχρονισμό της ε, προσέγγισης. Δηλαδή εννοώ ότι ε, η, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει την επεξεργασία της πρότασής της πολύ νωρίτερα από τη συζήτηση που έχουμε σήμερα. Το ερώτημα που θα ήθελα να σας θέσω. Είναι δυνατόν να συνεχίσουμε αυτή την αλακάρτ εφαρμογή διαφορετικών πολιτικών εάν επιθυμούμε μια καλύτερη ε, και πιο αποτελεσματική από διοικητικής απόψεως ε, ΚΑΠ. Ε, αναφερθήκατε επίσης στο ζήτημα της απλοποίησης και της ισότιμης κατανομής των επιδοτήσεων. Δεν θα πρέπει να δούμε και το ποιες είναι οι ιστορικές τιμές αναφοράς που λαμβάνουμε υπόψη μας και πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε τη σύγκληση, αν πραγματικά τελικά υπάρχει σύγκληση στο ιστορικό της Ένωσης. Πιστεύετε ότι αυτή η προσέγγιση με τις αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις είναι ενδεδειγμένη σήμερα όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Μήπως τελικά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία πιο δυναμικά, πιο, πιο στοχευμένα, πιο προσαρμοσμένα, έτσι ώστε τελικά να εγγεώμαστε το εισόδημα των γεωργών. Αυτά από πλευρά μου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εμένα μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Έχει πολλά θετικά στοιχεία. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση, γιατί μας είπατε ότι οι πληρωμές ε, παρουσιάζουν πολύ διαφορετικό ε, πεδίο, σε διαφορετική εικόνα σε διάφορα κράτη-μέλη. Αυτό έχει να κάνει με τη διατύπωση των αιτημάτων για την, ε, και των αξιώσεων για την ε, ενίσχυση ή με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εκμετάλλευση και η καλλιέργεια της γης. Και επίσης η επίτευξη των στόχων ή η ελλειπής επίτευξη καλύτερα μπορεί να οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο διατυπώνονται αυτά τα αιτήματα για τις ενισχύσεις. Γιατί φαντάζομαι ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιοι οποίοι δεν καλλιεργούν πράγματι τη γη. Και ίσως αυτό σχετίζεται και με το ιστορικό μοντέλο και τις ιστορικές τιμές αναφοράς. Άρα το μοντέλο πάνω στο οποίο έχουμε στηριχθεί για τους υπολογισμούς μας το 2000, τα τελευταία 18 χρόνια έχει βέβαια αλλάξει. Και είναι άλλοι αυτοί οι οποίοι τώρα πράγματι ε, εκμεταλλεύονται, καλλιεργούν τη γη. Κύριε Σουλαζό. Ευχαριστώ. Ζητήθηκε από την Επιτροπή να μας αναλύσει πώς μπορούμε να έχουμε και μία έτσι απλοποίηση του συστήματος και πώς μπορούμε να έχουμε ε, ουσιαστικό εισόδημα για τους γεωργούς για να συμβεί αυτό, νομίζω η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Χρειάζεται οι τιμέ τη αγορά, τι οποίε πολλούν τα προϊόντα του, οι αγρότε να είναι σωστέ, έτσι ώστε να μπορούν να ζήσουν από αυτέ και όχι τόσο από τι επιδιωτήσει, να μην βασίζονται στι υποδοτήσει. Και δυστυχώ αυτό δεν συμβαίνει. Και το πρόβλημα έγκυται και στου κανόνε. Θα σα μιλήσω για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ε, για το σιτάρι, α πούμε, στη Γαλλία, που το 1991 οι τιμέ ήταν πολύ υψηλότερε από, το ήταν στι τάξεις του 230 ε, ευρώ τον, τον, τόνο, ενώ τώρα έχουμε πέσει 149. Βλέπετε δηλαδή ότι πρόκειται για υποδιπλασιασμό σχεδόν. Και αυτό δημιουργεί ένα έλλειμμα. Ε, ε, έχουμε φτάσει, στο, οι αγρότες να πουλούν κάτω του κόστους, όταν το κόστος εκτιμούμε γύρω στο 170 ευρώ ανά τόνο. Και μην ξεχνούμε ότι οι φόροι δεν σταμάτησαν και τα υπόλοιπα τέλη να αυξάνονται. Επομένω, κατά την άποψή μα. δεν θα έπρεπε τα κυρίαρχα κράτη, μέλη, να, υποβάλουν, να επιβάλλουν στις χρηματαγορές ελάχιστες τιμές, κάτι που σήμερα απαγορεύεται. Επίσης έχουμε τις ε, περιοχές οι οποίες είναι λιγότερο αναπτυγμένες και οι οποίες ε, εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τις επιδοτήσεις. Είναι, είναι καταστροφική η αγροτική πολιτική γιατί είναι ισχύ αυτή την εξάρτηση από τις ειδικέ επιδοτήσεις. Εδώ δεν βλέπω ουσιαστικέ προτάσεις, έτσι ώστε τελικά να μειώσουμε την εξάρτηση των αγροτών από τις ε, επιδοτήσεις. Ε, σε αυτά τα ζητήματα, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να εστιάσουμε. Σας ευχαριστώ. Ο Χόισλινγκ. Ευχαριστώ πολύ για την έκθεση, αλλά δεν άκουσα μία λέξη. Τη λέξη περιβάλλον. Είτε στην επιτέξη των στόχων, γιατί η μεταρρύθμιση Τσόλος ήταν ε, υπό την ε, αιγίδα των καλύτερων επιδοτήσεων ε, προσφοράς στο κοινό, στο κοινό όφελο, στη βιοποικιλότητα το περιβάλλον. Αυτά δεν τα έχουμε καταφέρει. Αναφέρατε ωστόσο ενδιαφέροντα θέματα και επισημαίνω και αυτό εξ αρχής που μας είχαν απασχολήσει στην προηγούμενη μεταρρύθμιση και ένα από αυτά ήταν η δυνατότητα για απλοποίηση με τους στόχους που ορίζουμε και αν μπορούν οι ενισχύσεις να καταβάλλονται χωρίς διαφοροποίηση με μέτρο το εκτάριο. Βεβαίως, με μέτρο το εκτάριο θα ε, εποφεληθούν περισσότερο μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό προκύπτει και με την προηγούμενη αλλά και με την τωρινή ΚΑΠ. Και συνεχίζεται γιατί οι μεγαλύτερες είναι αυτές οι επιχειρήσεις οι οποίες επωφελούνται από τις ε, ενισχύσεις. Άρα δεν έχει ρυθμίσει το ζήτημα. Μήπως έπρεπε να μας πείτε λοιπόν για να λυθεί αυτό το ένιγμα ποια μέτρα, ε, ποια κριτήρια θα έπρεπε να ακολουθήσουμε. Και επίσης τι χρειάζεται συγκεκριμένα ο Γεωργός. Χρειάζεται υποστήριξη στο εισόδημά του εάν έχει ένα συμπληρωματικό εισόδημα και δεν εξαρτάται από τη γεωργική του δραστηριότητα, ξεκολουθεί να, χρειάζεται την ενίσχυση. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα κοιτάξουμε, να αναζητήσουμε τι, ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες του δικαιούχου. Και είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί μεγάλες διαφορές βλέπουμε και μέσα στην ίδια εκμετάλλευση. Κάποιοι που με χαμηλές τιμές ακόμη μπορούν να έχουν καλό προϊόν και καλή λειτουργία στην εκμετάλλευσή τους, κάποιοι που δεν τα καταφέρνουν. Φερρυπίν. Η αποσύνδεση. Είναι η μόνη χώρα η Γερμανία, από ό,τι γνωρίζω, η οποία έχει προχωρήσει σε πλήρη αποσύνδεση, με πολλά μειονεκτήματα, κατά το δικό μου κριτήριο. Δεν υποστηρίζω την πλήρη αποσύνδεση, διότι στη Γερμανία, επί παραδείγματι, έχουν πληγεί ιδιαιτέρως οι ε, κτηνοτρόφοι προβάτων, εγωπροβάτων που δεν ε, μπορούν να λάβουν ενίσχυση αναέκταση, αναεκτάριο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να ξανακοιτάξουμε δηλαδή. Αλλά μια και ανέφερε την γαλακτοπαραγωγή ο Άλμπερτ Ντες, η οποία εξαρτάται τόσο πολύ από τις ε, ενισχύσεις για το γάλα. Ε, δεν νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το εξαντλήσουμε σε μια τέτοια διαπίστωση. Υπάρχει μια προϊστορία και η προϊστορία είναι η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς πρέπει να μα ξαφνιάζει λοιπόν, αφού θελήσαμε την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς, το γεγονός ότι έχουμε φτάσει στα 60 ε, λεπτά του ευρώ στο λίτρο του γάλακτος. Δεν μπορεί βεβαίω να επιβιώσει κανένα γαλακτοπαραγωγό. Βεβαίω χρειάζονται μηχανισμοί στην αγορά και παρεμβάσει οι οποίε να ρυθμίζουν τι τιμέ. Δεν μπορούμε να αφήσουμε απόλυτη ε, ελευθερία στην ε, αγορά, άκρατη ελευθερία στην αγορά σε βαθμό που για τις επόμενες δεκαετίες να εξαρτάται ο γαλακτοπαραγωγός από την ενίσχυση. Θα ήθελα και σε αυτό να πείτε δύο λόγια. Και τελευταία κουβέντα. Για το μέλλον και από αυτά που μας έχει πει ο Επίτροπος για τη μελλοντική γεωργική πολιτική πάλι διαπιστώνω ότι δεν ε, θα είναι δυνατή η υλοποίηση των στόχων πάλι με την απελευθέρωση και πάλι με ε, μια παρεπίπτουσα αναφορά στο ότι θα πρέπει να κάνουμε πράγματα που να είναι υποφέλη για το περιβάλλον. Δεν εξυπηρετούμε έτσι τους στόχους μας, προχωρούμε σε μια άκρατη απελευθέρωση και δεν μπορούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και τη γεωργία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σένερα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και το Ανεκτικό Συνέδριο για την έκθεσή του. Μήπως θα μπορούσατε να μας κάνετε μια πιο αναλυτική αναφορά των θεμάτων της σύγκλησης. Γιατί μας είπατε στην έκθεση ότι οι ενισχύσεις ε, ευνοούν κυρίως τις μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν, είναι βιώσιμο ένα γεωργικό σύστημα όπου οι μεγάλες ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή εγκαταστάσεις ε, χρειάζονται δημόσιες ενισχύσεις για να επιβιώσουν. Γιατί αν ε, ε, στη Γεωργία θέλω να είμαστε ανταγωνιστικοί, αλλά μόνο οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις, ε, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι ανταγωνιστικές και τη συνέχεια επεκτείνονται, πώς αυτές είναι, αυτές που κατεξοχήν επιδοτούνται για να επιβιώσουν. Θα πρέπει να αναλύσουμε νομίζω πιο διεξοδικά αυτό το θέμα. Επίσης, θα ήθελα να μου παρουσιάσετε πιο αναλυτικά τα πορίσματά σας για την ανισορροπία μεταξύ των ε, μικρών γεωργών ε, από τις διάφορες πολιτικές και μάλιστα ολόκληρο τομείς μερικές φορές έχουν αποκλειστεί από τη λήψη ενισχύσεων. Επίσης κάνετε μια εκτίμηση της ανισότητας που υπάρχει σε ό,τι αφορά την ε, λήψη των ενισχύσεων από τις γυναίκες κυρίως, Γιώργος, από τις αγρότησες. Ευχαριστώ κύριε Αγγιλέρα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου για την έκθεση που μας υπέβαλε. Ενδιαφέρουσα η ανάλυση που κάνει το Ελεκτικό Συνέδριο για τις βασικές ενισχύσεις και τον αντίκτυπο που έχουν αυτές. Επίσης κάνετε μια αξιολόγηση των μέτρων τη στιγμή που εφαρμόζεται η κυνηγιορική πολιτική. Αλλά νομίζω ότι έχουμε ελάχιστα στοιχεία στη διάθεσή μας. Το αναφέρατε και εσείς κάπου. Αλλά έχουμε και κάποια στοιχεία που είναι δύσκολο να αξιολογηθούν. Γιατί η περίοδος 2013-2020 ε, και τα μέτρα της άρχισαν να εφαρμόζονται καθυστερημένα από τα κράτη-μέλη. Και μόνο δύο χρόνια, σε δύο, για δύο χρόνια είχε εφαρμοστεί ε, το καθεστώς βασικών ενισχύσεων. Οπότε είναι δύσκολο να αξιολογήσουμε τα στοιχεία από την μεταρρύθμιση αυτή, αν δεν πάρουμε μια μεγαλύτερη χρονική απόσταση. Μπορούμε να δούμε κάποια τάση ίσως, κάποια κατεύθυνση, αλλά τα στοιχεία που είδα στην έκθεσή σας τουλάχιστον αφορούν το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και την κοινή γεωργική πολιτική σε προηγούμενες περιόδους. Γιατί για την τωρινή περίοδο 2013-2020 είναι πολύ πρόημο να αξιολογήσουμε μέτρα όπως το greening, την οικολογικοποίηση και άλλα μέτρα. Ένα άλλο εντυπωσιακό σημείο ε, το οποίο θα ήθελα να μου αναλύσετε είναι το εξή. Αναγνωρίζετε ότι η ΚΑΠ συνέβαλε ή βοήθησε στην εδαφική συνοχή. Δηλαδή μείωσε τις ε, εισοδηματικές διαφορές ε, των αγροτικών τι αστικές περιοχές, τη διαφορά στο κατακεφάλαιο εισόδημα. Οπότε η ανισότητα μειώθηκε, είπατε, γιατί αυτό συμβάλλει πραγματικά στην εδαφική συνοχή. Έχετε όμω πιο διεξοδικά στοιχεία για να ε, τεκμηριώσετε αυτή τη διαπίστωση που ήταν ενδιαφέρουσα. Επίσης, ε, είναι περίπλοκο στο ισχύον σύστημα ε, να γίνει μια αξιολόγηση γιατί χορηγούνται τα κονδύλια στα κράτη πρώτα και μετά εγκρίνονται τα μέτρα, ιδιαίτερα στο δεύτερο πυλώνα. Και στη συνέχεια κάθε χώρα επιλέγει τι θα εφαρμόσει από τον πρώτο πυλώνα. Τώρα, με την αλλαγή που εσείς κρίνετε θετική, με την υποβολή των στρατηγικών σχεδίων δράσης, θεωρείτε ότι αυτό θα είναι το, το κλειδί της ε, επιτυχής μελλοντικής ΚΑΠ, τα στρατηγικά σχέδια. Δηλαδή, πρώτα θα πρέπει να βλέπουμε τα αποτελέσματα και μετά να καταβάλουμε τι ενισχύσει. Να περιμένουμε πρώτα να δούμε αποτελέσματα και μετά να πληρώνουμε. Αυτό έρχεται σε αντίφαση με το πρώτο πυλώνα. Μπορεί να λειτουργεί για το δεύτερο πυλώνα, αλλά όχι για το πρώτο. Με αυτέ τι παρατηρήσει ε, θα ήθελα παρόλα αυτά να σα συγχαρώ, γιατί θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρουσα η δική σα έκθεση και θα ε, κριθεί χρήσιμη για την περαιτέρω συζήτηση. Κυρία Χόιμπουχ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την έκθεση. Δεν μας ξαφνιάζει το συμπέρασμα ότι υποφελούνται περισσότερο οι μεγάλες επιχειρήσεις, βεβαίως. Εφόσον ε, ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις ε, γεωργικές εκτάσεις, όποιος έχει μεγαλύτερη έκταση υποφελείται περισσότερο. Λογικό είναι. Ωστόσο, με ξαφνιάζει το ότι ε, ίσως μπορείτε να κάνετε κάποιες προτάσεις για πολιτικούς στόχους. Σας έχει απασχολήσει αυτό, ποιος θα είναι ο κύριος στόχος, ο γενικός καλύτερα στόχος και μετά οι επιμέρους συγκεκριμένοι στόχοι. Θα πρέπει να συζητήσουμε Φερρυπίν, στο στόχο προστασίας του περιβάλλοντος. Θα αρκούσε να πούμε θέλουμε να περιορίσουμε την χρήση των ζεζανιοκτώνων Ή θα έπρεπε να βρούμε μια διαφορετική διατύπωση. Πώς θα έπρεπε να διατυπωθούν αυτοί οι στόχοι. Επίσης η ενίσχυση ανάλογα με τις ανάγκες, τις πραγματικές του κάθε γεωργού που ανέφερε ο κύριος Χόισλινγκ. Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η πρόταση. Πώς όμως μπορούμε να την υλοποιήσουμε και πώς, έχοντας διατυπώσει στόχους, φερρυπίν περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, ε, τι κάνουμε, ενισχύουμε τον στόχο ή ενισχύουμε την ανάγκη ε, του γεωργού, την οικονομική ανάγκη του γεωργού. Πώς θα μπορούσαμε να το διατυπώσουμε αυτό και στο θέμα της αγοράς. Εάν χάνουμε μόνο στη Γερμανία 10 λεπτά του ευρώ στο γάλα, σημαίνει ότι χάνουμε 3,2 δις χρήματα σε ευρώ πάντα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Άρα είτε αποτυγχάνει η αγορά στην ελεύθερη αυτή λειτουργία, είτε δεν αντέχουν, δυστυχώς πρέπει να το πούμε, οι γαλακτοπαραγωγικές μονάδες τον ανταγωνισμό. Εδώ νομίζω ότι δεν μπορούμε με τις άμεσες ενισχύσεις να κάνουμε την αντιστάθμιση. Θα πρέπει να κάνουμε δράσεις απευθείας στην αγορά για να αποκαταστήσουμε τις συνθήκες ε, λειτουργίας και πώλησης. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα συγκεκριμένα να μας πείτε τι μέτρα θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε και με ποιους στόχους, ε, με ποιους στόχους, ποιους στόχους θα έπρεπε να ορίσουμε για να μπορούμε να κάνουμε την επαλήθευση ότι υλοποιήθηκαν. Κυρία Ράνς Καρσία, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Φιγκερέδο, το μέλος του Ελεκτικού Συνεδρίου για την υποβολή της ειδική αυτής έκθεσης. Ψάχνετε, εδώ είμαι. Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή την παρουσίαση και διάβασα την έκθεση που μιλάει για περιορισμένη, περιορισμένο αντίκτυπο στη σύγκληση. αλλά θα ήθελα να επικεντρωθούμε περισσότερο στην απλούστευση. Την περασμένη, το περασμένο Σαββατοκυριακό είχα μια συνάντηση με γεωργού που μου επισήμαναν ότι το μείζον πρόβλημα τη κοινή γεωργική πολιτική είναι ότι κάθε φορά που την απλοποιούμε, την καθιστούμε πιο περίπλοκη. Νομίζω ότι ο πρωταρχικό στόχος είναι να είναι προσβάσιμη, προσιτή η κοινή γεωργική πολιτική για τους γεωργού και με τους ελέγχους φυσικά που είναι απαραίτητοι. Θα πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε περισσότερο στο ρόλο της απλούστευσης. Έχουμε όλα τα τεχνικά μέσα στη διάθεσή μας για να το επιτύχουμε. Θα πρέπει όμως να δείξουμε μεγαλύτερη ευαισθησία απέναντι στου γεωργού και στα μέσα που διαθέτουν οι γεωργικοί κτηνοτρόφοι, που είναι και οι βασικοί αποδέκτε τη κοινή γεωργική πολιτική. Ο κ. Ντόρφμαν μα είπε ότι θα είναι δύσκολο να καταλήψουμε το ιστορικό μοντέλο, τουλάχιστον μερικέ χώρε μέλη. Μιλήσαμε για το ρόλο του ενεργού αγρότη. Θα ε, ήθελα όμω να επικεντρωθούμε στα αποτελέσματα. Ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα θα ήταν από την εφαρμογή τη κοινή γεωργική πολιτική είναι να μετρήσουμε το επίπεδο τη ηλικιακή ανανέωση ε, των Ευρωπαίων Γεωργών και Κτηνοτρόφων, γιατί εκεί έχουμε μεγάλη, μεγάλο πρόβλημα στην ανανέωση των γενεών η μέση ηλικία του γεωργού και κτηνοτρόφου είναι ανησυχητική. Γιατί υπάρχει γύρανση και του γεωργικού πληθυσμού και του κτηνοτροφικού πληθυσμού. Δεν υπάρχει ηλικιακή ανανέωση στη γεωργία και την κτηνοτροφία για να επιτρέψουν την διατήρηση τη κοινή γεωργική μα πολιτική. Εσεί πώ βλέπετε στο ελεκτικό συνέδριο τι προσπάθειε που κάνουμε να βοηθήσουμε του νεαρού αγρότε στον πρώτο και δεύτερο πυλώνα. Οι στόχοι που θέσαμε έχουν αποφέρει καρπούς. Και ω προ την απασχόληση, μα είπατε ότι μεγάλε γεωργικέ εκμεταλλεύσει ε, δέχονται τα περισσότερα κονδύλια. Τι επίπεδο απασχόληση όμω ε, εξασφαλίζουν, γιατί έχουμε οικογένειε ε, του γεωργικού κλάδου που αποφελούνται από αυτό ή αυτοαπασχολούμενους που απασχολούνται σε τέτοιες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Τι θέσεις απασχόλησης δημιουργούν αυτές οι μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και έχουν κάποιο κοινωνικό αντίκτυπο, γιατί είναι μεν λαμβάνουν τα περισσότερα κονδύλια, αλλά παρουσιάζουν και κάποιο έργο προ την απασχόληση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Φιγκερέντο, τον εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου για την υποβολή της έκθεσης που δείχνει ότι σε πολλούς τομείς θα πρέπει να κάνουμε κάποιες βελτιώσεις και ίσως θα πρέπει να πάμε επί τόπου να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει στους αγρούς, στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Γιατί ίσως έχουμε μια πολύ θεωρητική εντύπωση για τη γεωργία. Μερικές μικρότερες φάρμες, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, έχουν κληρονομηθεί στους τωρινούς δικαιούχους, ενώ ε, σε άλλες ε, οι ιδιοκτήτες χρειάστηκε να δανειστούν για να ξεκινήσουν η ορική δραστηριότητα. Αν θέλουμε να μεταρρυθμίσουμε την ΚΑΠ, θα πρέπει ε, η μεταρρύθμιση να στοχεύει στην απλούστευση, γιατί παρά είναι περίπλοκη σήμερα εκείνη η γεωργική πολιτική. Αυτό που μου λείπει είναι η καλύτερη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη γεωργία ώστε να έχουμε βοήθεια και ενίσχυση, αλλά και καλύτερη αξιοποίηση και εφαρμογή της τεχνολογίας, γιατί εκεί υπάρχουν μεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα. Και Επίσης, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι διαφορετικές από τη χρήση σουλφιτών, θείουχων ενώσεων φυτοφαρμάκων. Δίνονται βασικές ενισχύσεις ε, στρεματικές, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε διαφάνεια, απλοποίηση και δικαιοσύνη ισοτιμία στην ε, εφαρμογή της κοινή γεωρικής πολιτικής. Και αν κάνουμε διάκριση μεταξύ των μεγάλων και μικρών γεωρικών εκμεταλλεύσεων, Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει άνηση κατανομή. Ίσως θα πρέπει τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις να τις κατακαιρματίσουμε σε μικρότερες για να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ομοιομορφία στην κατανομή. Στόχος πάντως είναι η απλούστευση. Και να δούμε και την κατάσταση ανά χώρα Έχοντα όμω κατά νου και τις παγκόσμιες τιμέ αγορά, γιατί εκεί ανταγωνιζόμαστε, στην παγκόσμια αγορά. Οπότε δεν μπορούμε να διαφορούμε, να για τις παγκόσμιες τιμέ. Θέλουμε λοιπόν και να ευνοήσουμε τους γεωργού και να καταστήσουμε πιο απλή την κοινή γεωργική πολιτική. Κάτι που αποτελεί δύσκολο φυσικά έργο. Επίση, αν δούμε την επιδημία τη Αφρικανική Πανόλη των χείρων και πώ επηρέασε την Ευρώπη, μερικές χώρες κατάφεραν να περιορίσουν την έκθεση στην επιδημία και άλλες όχι. Ίσως αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει προϋπόθεση για τη λήψη των ενισχύσεων. Κύριε Μιούλερ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου για την πολύ διεξοδική αυτή παρουσίαση. Ήταν σωστή η επιλογή της ενίσχυσης των γεωργών. Οι εθνικές αρχές έχουν κάποιες δυσκολίες αντιμετωπίσει κατά την υλοποίηση, το αντιλαμβάνομαι και εγώ. Θα ήθελα ωστόσο να επισημάνω ότι μου προξένησε μια κάποια δυσφορία το γεγονός που αναφέρεται στην έκθεση ότι σε κάποιες χώρες όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμα και η Ελλάδα έχουν μόνο κατεκτήμηση υπολογισμού ή προσωρινούς υπολογισμού, Κάτι το οποίο εμένα για τη Γερμανία μου φαίνεται αδιανόητο, γιατί έχουμε κάθε ε, κομμάτι γης, κάθε θάμνο, κάθε φράχτη τους έχουμε υπολογίσει, καταγράψει και συμπεριλάβει στον υπολογισμό των ενισχύσεων. Γιατί λοιπόν να καθυστερούν κάποια κρατημέλη στη συλλογή των δεδομένων που απαιτούνται για την επακριβή ε, καταγραφή των εκτάσεων. Υπάρχει το σύστημα GPS που διευκολύνει τόσο πολύ αυτό το έργο. Και επίσης θα ήταν καλό να λάβουμε υπόψη και φέτος ε, αυτά που μπόρεσαν να λυθούν σε σχέση με τον κανονισμό Omnibus ως προς την έννοια του ενεργού γεωργού και επίσης εκεί που η Επιτροπή θέλει με παράγοντες να δώσει απαντήσεις στην ανάλυση επί παραδείγματι του δημοσίου αγαθού και που οι συνάδελφοι θέλησαν να θέσουν στην επιχειρηματολογία ως ένα μέρος της, του υπολογισμού του, κέντρου, του κέρδους ε, ε, εάν απαγορευτεί ένα μέρος της ε, εντατικής παραγωγής και αφαιρεθούν κάποια χρήματα από τις μεγάλες επιχειρήσεις, παραδείγματι. γιατί η Επιτροπή μας έχει πει ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν περί το 72% των συνολικών ενισχύσεων, αλλά από την άλλη κλιματική αλλαγή τι σημαίνει, οι στόχοι για το κλίμα τι σημαίνει, ε, η ε, εκτροφή αγελάδας ξέρουμε ότι ε, οδηγεί σε παραγωγή μεθανίου. Σε ποιο βαθμό αυτό ανατρέπει την υλοποίηση των στόχων για την κλιματική αλλαγή. Νομίζω ότι μπορούμε και με την αποσύνδεση στις άμεσες αυτές ενισχύσεις να δώσουμε κάποια καλά αποτελέσματα και για τις ε, μεγάλες αλλά και για τις εκτατικές εκμεταλλεύσεις. Θα ήθελα λοιπόν πιο συγκεκριμένες ιδέες ως προς τους παράγοντες που μπορεί η Επιτροπή να αξιοποιήσει για την ανάλυση της έννοιας του δημοσίου αγαθού. Και ούτω ή άλλω νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία και στο προσεχέ θέμα τη ημερησία διάταξη να δούμε τι ιδέε αυτέ σε λεπτομέρεια. Eh, Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για το ελεγκτικό συνέδριο για την εξαιρετική ποιότητα έκθεση. Αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα είναι ότι οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις είναι αυτές που κερδίζουν περισσότερο. Έχουμε αριθμητικά στοιχεία στη διάθεσή μας. Είναι προφανές. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχω θέσει πολλές φορές. Εγώ είμαι υπέρ των μικρών οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, γιατί αυτές είναι που θα διασφαλίσουν την επιβίωση το, της περιφέρειας. Το ερώτημα είναι τι είδους ε, Ευρώπη θέλουμε στο μέλλον, σε τι είδους Ευρώπη θα θέλουμε να ζούμε. Ε, και για να το απαντήσουμε αυτό θα πρέπει να δούμε σε ποιες συνθήκες διαβιούν οι αγρότες. Πρέπει να διασφαλίσουμε το αγροτικό εισόδημα, έτσι ώστε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουν να ζουν και να καλλιεργούν τη γη τους. Επηρεάζονται βεβαίω από κανονισμού που σάγουμε για παράδειγμα γιατί τα νητρικά και για τα λοιπάσματα, αλλά η κλιματική αλλαγή είπαμε ότι κατά κύριο λόγο θα καταπολεμηθεί με τη μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. Επομένω θα πρέπει να δούμε μέτρα τα οποία να βοηθούν ιδιαίτερα τις μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και όχι τις μεγάλες επιχειρήσεις. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να πηγαίνουμε προς τα εκεί. Επίσης, τίθεται και το ε, ερώτημα της ε, βοήθειας που δίνουμε στους πολίτες που έχουν ε, μεγαλύτερη ανάγκη στις χώρες μας. Γιατί πολλοί συνάδελφοι αναφερθήκαν σε αυτές τις επιδοτήσεις και είπαν «Μα είναι τόσο μεγάλες». Πώς όμως τελικά το ποσοστό αυτών των επιδοτήσεων φτάνει στους ίδιους τους αγρότες και πόσο φτάνει σε εκείνους που ίσως είναι ε, ιεραρχικά οι ανώτεροι σε αυτούς σε μια μεγάλη επιχείρηση που τους πεταλεύεται. Ε, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η έκθεση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Βεβαίως συζητούμε αυτή τη στιγμή για την κοινή αγροτική πολιτική και θα είναι αναπόφευκτο να υπάρξει μια κάποια μείωση εξαιτία του Brexit. Είναι προφανές ότι θα υπάρχουν λιγότεροι διαθέσιμοι πόροι. Και υπάρχουν και άλλες πιέσεις για χρηματοδότηση άλλων τομέων, πέραν δηλαδή της γεωργίας. Και λέγεται ότι χρειάζεται να διασφαλίσουμε την αγροτική παραγωγή και την διατροφική μας ασφάλεια και για αυτό πρέπει να το πράξουμε μέσω μιας ισχυρής κάπου. Διαπιστώνουμε όμω ότι δεν έχουμε ουσιαστική σύγκληση. Ότι δεν έχει προχωρήσει η στόχευση. Ότι δεν έχει προχωρήσει η απλοποίηση. Και με αυτόν τον τρόπο γίνεται ακόμα πιο δυσχερέστερο σε εμά να παρουσιάσουμε και να πουλήσουμε, αν θέλετε, την κοινή αγροτική πολιτική στο κοινό, στου πολίτε. Αυτό που θέλω εγώ να μπορώ να πω στου πολίτε μου είναι ότι τα αξιοποιούμε αυτά τα χρήματα ε, ε, προ το κοινό καλό. Όχι να μπορούν να μου ανταπαντήσουν ότι υπάρχουν οι οποίοι υποφελούνται υπερβολικά ή ακόμα και ορισμένοι οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτά τα χρήματα όχι για να βοηθήσουν το αγρόκτημά τους, αλλά για να αγοράσουν ε, προϊόντα πολυτελείας. Και το ερώτημά μου είναι το εξής. Δεν πιστεύετε ότι είναι πιο δύσκολο για εμάς να παλέψουμε, να κρατήσουμε την κοινή αγροτική πολιτική στο επίπεδο που έχει και ακόμα μεγαλύτερο, αν θέλετε, ακριβώς το γεγονός αυτό ότι δεν, έχουμε, ε, ότι δεν έχουμε σύγκληση και ότι τα χρήματα δεν φτάνουν στους δικαιούχους που θα έπρεπε. Δεν είναι κάτι, ένα στοιχείο αυτό το οποίο μας δυσχεραίνει εμάς που θέλουμε να υπερασπιστούμε τους αγρότες και το εισόδημά τους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπάσκο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Φιγερέρο που μας δίνετε και αυτή τη δυνατότητα να συζητήσουμε την έκθεση την ειδική του ελεκτικού συνεδρίου για το βασικό ε, σύστημα ενισχύσεων. Πρώτα απ' όλα, να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει την έκθεση. Λαμβάνουμε υπόψη μας όλες τις συστάσεις που απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις έχουμε αποδεχθεί όλες. Βεβαίως, δεν θα μπορούσα να προκαταλάβω αυτή τη στιγμή με ποιον τρόπο συγκεκριμένα ε, θα τις εκφράσουμε αυτές τις ε, συστάσεις, θα φροντίσουμε να υλοποιηθούν αυτές τις συστάσεις μέσω των συγκεκριμένων νομοθετικών μας προτάσεων το 2020. Χαίρομαι ότι το γενικό συμπέρασμα της έκθεσης ε, για το βασικό σύστημα ενίσχυσης είναι θετικό. Ο βασικός στόχος ήταν να διασφαλίζεται το αγροτικό εισόδημα και έχουμε μια δαπάνη της τάξης των 18 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο για να γίνεται αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, ε, βοηθήσει τα κράτη-μέλη να εισαγάγουν αυτό το σύστημα, να το υλοποιήσουν και το παρακολουθεί την εφαρμογή του. Επομένως έχει εμπλακεί και στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή και στην παρακολούθηση. και όπως αναφέρει και το ελεγκτικό συνέδριο, η εφαρμογή του συστήματος των βασικών ενισχύσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εθνικές αρχές. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο αφορά 4 εκατομμύρια αγρότες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και διαπιστώνουμε ότι η χρήση των κονδυλίων αυτών δεν οδήγησε σε ουσιώδη σφάλμα, σε κίνδυνο για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Επομένω, μπορούμε να πούμε ότι είναι επιτυχέ το σύστημα συνολικά. Βεβαίω, υπάρχουν κάποια στοιχεία που η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου μα επισημαίνει ω στοιχεία που πρέπει να βελτιωθούν, όπω για παράδειγμα η απλοποίηση ή το πριν. Και θα αναφερθώ πιο συγκεκριμένα στα τρία κύρια ζητήματα που μα επισημαίνει το Συμβούλιο. Ξεκινώντα από την απλοποίηση η αρχική πρόταση της Επιτροπής για την τρέχουσα περίοδο πολιτικής είχε λιγότερες επιλογές. Ωστόσο, μέσω της διαδικασίας της συναπόφασης, μέσω της ε, συνομοθέτησης της διαδικασίας αυτής, προσθέθηκαν και άλλες επιλογές, έτσι ώστε λεγόταν να είναι η πολιτική πιο ευέλικτη, να μπορεί να προσαρμοστεί στις εθνικές ιδιωτερότητες. Αυτό όμως οδηγεί και σε πιο περίπλοκους κανόνες. θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η αρχική πρόταση της Επιτροπής σε σχέση με τον ενεργό ε, ακρότη ήταν πολύ πιο περιορισμένη και συγκεκριμένη ε, από αυτό που τελικά είδαμε να εφαρμόζεται τα τελευταία 4-5 χρόνια. Όσον αφορά τη στόχευση. Σε ορισμένα κρατημέλη αποκλείστηκαν εκείνες οι εκμεταλλεύσεις οι οποίες έχουν μόνο σε μικρό βαθμό αγροτική ε, παραγωγή, στις στόχους τους και εδώ πιστεύω θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι να αναγνωρίσουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μεγάλος κατακαιρματισμός του αγροτικού τομέα, πάνω από 7.000, 7 ε, εκατομμύρια δικαιούχοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, δεν μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει όλες τις ιδιαιτερότητες ε, αυτών των εκμεταλλεύσεων χωρίς να δημιουργήσει ένα γραφειοκρατικό τέρας. Υπάρχουν και άλλα συστήματα υποβοήθησης, για παράδειγμα για τις μικρές εκμεταλλεύσεις, για τους νέους γεωργούς, η χρηματοδότηση για την οικολογικοποίηση και άλλα δηλαδή μέτρα και, άλλα, ε, και άλλοι τρόποι που μπορούμε να αξιοποιήσουμε το υφιστάμενο σύστημα για να βοηθήσουμε συγκεκριμένες ομάδες ε, γεωργών ή, συγκεκριμένου ή συγκεκριμένους άλλους στόχους πολιτικής. Και τέλος, το τρίτο θέμα που θέτει το ελεγκτικό συνέδριο και στο οποίο διαπιστώνει ε, καθυστέρηση στην πρόοδο είναι η σύγκληση. Γνωρίζετε ότι τα κράτη-μέλη είχαν τρει επιλογές, είτε, προσπαθ... είτε να επιδιώξουν γρήγορα τη σύγκληση, είτε προς το τέλος της προγραμματικής περίοδου, είτε, εάν ζητούσαν παρέκκληση, να επιδιώξουν μόνο μερική σύγκληση. Η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική από κράτος μέλος σε κράτος μέλος και έχουμε επίσης και μια περιφερειακή εφαρμογή αυτών των πολιτικών που έχει επιπτώσεις. Ωστόσο, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ο τελικός στόχος συμπεριελήφθη στην πρόταση την αρχική της Επιτροπής την Ομοθετική που ήταν ο τελικός στόχος να καταλήξουμε σε μία ενιαία επιδότηση σε ολόκληρη την, την, Ένωση. Όταν όμως συζητούμε αυτά τα τρία ζητήματα, της απλοποίησης, της σύγκλησης, της στόχευσης. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη δημοσιεύσει μια ανακοίνωση για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής, στο οποίο εξετάζει ε, μοντέλα και, και πιθανά σενάρια για το τι θα συμβεί μετά το 2020, επιδιώκοντας μέσω αυτής της συζήτησης να οδηγηθούμε σε ένα, σε ένα πλαίσιο πολιτικής το οποίο θα είναι απλούστερο, πιο στοχευμένο, και θα έχει μια προσέγγιση η οποία θα, θα βασίζεται περισσότερο στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Δεν θα μπω περισσότερε λεπτομέρειε βέβαια αυτή τη στιγμή γιατί θα έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μα στο άμεσο μέλλον να τα συζητήσουμε αυτά. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στις επισημάνσεις που κάνει το Ελεκτικό συνέδριο όσον αφορά την, τον υπολογισμού σε ορισμένα κράτη-μέλη. Ε, συμπίπτουν τα ευρήματα του Ελεκτικού συνεδρίου με αυτά τη επιτροπή. Και μετά από οποιοδήποτε τέτοιο εύρημα έχουν ξεκινήσει οι σχετικές διαδικασίε ε, στο, στο πλαίσιο της συμμόρφωση. Θεωρεί το Ελεκτικό συνέδριο ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των οργανισμών πιστοποίησης. Και εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί. Οι οργανισμοί πιστοποίηση είναι εκείνοι οι οποίοι θα πρέπει να διεξάγουν του ελέγχου και αυτό είναι κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα και το προωθεί η Επιτροπή μέσω των κατευθυντηρίων γραμμών τη. Ε, Σημερασματικά θα έλεγα ότι υιοθετούμε όλε τι προτάσει του ελεκτικού συνεδρίου, τι συστάσει μάλλον του ελεκτικού συνεδρίου και ήδη έχουμε ξεκινήσει να, ε, να προσπαθούμε για την πλήρη εφαρμογή του. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Διευθυντά. Ο κύριος Φλάναγκαλ θέλει το λόγο για περώτηση. Συγγνώμη, μια σύντομη ερώτηση. Μας είπατε ότι έχουμε τρία διαφορετικά συστήματα που εφαρμόζονται στην Ευρώπη. Όντως, είναι πολύ διαφορετικά αυτά τα τρία συστήματα. Α, όμως, η γεωρική πολιτική λέγεται κοινή γεωρική πολιτική πού έγινε το κοινό της γεωργικής πολιτικής. Μήπως θα πρέπει να αλλάξουμε την, τον τίτλο της, γιατί δεν νομίζω ότι ανταποκρίνεται το περιεχόμενο στον όρο. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε την υποβολή των ερωτήσεων. Ε, παρατάθηκε αυτή, αυτό το τμήμα της συνεδρίασης, αλλά ήρθε η ώρα για τις απαντήσεις και με μεγάλη χαρά θα δώσω το λόγο στον κύριο Φιγκερέντο για να απαντήσει στους ευρωβουλευτές, παρακαλώ. Επ' ευκαιρία να καλωσορίσω και τους καλεσμένους κυρίας Μίλλερ από τη Βαβαρία. Καλώς ήρθατε. Έχετε πολύ καλή εκπροσώπηση στην Επιτροπή Γεωργίας. Σας ε, καλωσορίζουμε εγκάρδια. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου ξαναδίνετε το λόγο. Και ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας για τις πολυάριθμες ερωτήσεις τους. Ήταν τέτοιος ο καταιγισμός των ερωτήσεων και μάλιστα καλύπτουν ένα τόσο ευρύ φάσμα που φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω να απαντήσω σε όλες. Γιατί ακριβώς οι ερωτήσεις σας αντικατοπτρίζουν, και φοβάμαι ότι θα συμφωνείτε μαζί του, αντικατοπτρίζουν το πόσο δύσκολη είναι η συζήτηση. Η κοινή γεωρική πολιτική είναι η αρχαιότερη κοινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει μακρά ιστορία και χειρίζεται σημαντικά δημόσια κονδύλια και επίσης ε, συνδέεται με την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με σημαντικά θέματα τα τρόφιμα για τους Ευρωπαίους, την επιστηστική ασφάλεια των Ευρωπαίων και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα επιμέρους θέματα καθιστούν ιδιαίτερα περίπλοκη και σύνδετη συζήτηση. Και πολλές από τις ερωτήσεις σας φοβάμαι ότι περισσότερο έχουν να κάνουν με το μέλλον της ΚΑΠ παρά με το παρελθόν. Θα διαμορφώσουν την νέα, τη μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική παρά το ισχύον σύστημα ε, του βασικών ενισχύσεων προς τους γεωργούς. Και περισσότερο προβληματίζονται για το μέλλον και προβληματίζουν για το μέλλον όλες αυτές οι ερωτήσεις που υποβάλλατε. Εμείς στην ειδική έκθεση για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης που σας παρουσίασα, πούμε ότι γενικώ το σύστημα είναι σε καλό δρόμο, αυτό που εννοούμε είναι ότι υπογραμμίζουμε κάποια σημεία και σας ευχηστούμε την προσοχή σε αυτά. Θα ήθελα να επικεντρωθείτε στα σημεία που αναφέρομαι στην έκθεσή μας και που αφορούν όχι μόνο την απλοποίηση, αν και η απλοποίηση είναι επίσης σημαντικό θέμα, αλλά αφορούν τη σύγκληση που επίσης είναι σημαντικό θέμα και κατά τη γνώμη μου αφορούν το πιο σημαντικό θέμα, τη στόχευση. Ερωτώ λοιπόν, τα κονδύλια που αφιερώνουμε στην κοινή γεωργική πολιτική φτάνουν στα χέρια των γεωργών που πραγματικά τα χρειάζονται. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα που αναλύει ο δημοσιονομικός ελεγκτής. Και ως τέτοιος ελεγκτής θα έλεγα ότι μετά από ανάλυση των ερωτήσεων καταλήγουμε σε 8 κύρια προβλήματα. Και αυτά προκύπτουν από τις δικές ερωτήσεις και απορίες. Το πρώτο μείζον πρόβλημα είναι το θέμα της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη γεωργία. Δεν χρησιμοποιήσετε ακριβώ αυτούς τους όρους, αλλά πολύ μιλήσατε για τους στόχους, για το αντικείμενο, για τους σκοπούς, τους στόχους της ευρωπαϊκής ε, κοινής γεωργικής πολιτικής. Και αυτός θα είναι και ο βασικός προβληματισμός του νομοθέτη για τη μελλοντική ΚΑΠ. Ποιοι είναι οι στόχοι της κοινή γεωργικής πολιτικής ποιους στόχους θέλουμε να υλοποιήσουμε με την κοινή πολιτική. Αυτό είναι το μείζον ερώτημα. Γιατί αν δεν είμαστε σαφείς ως προς τους στόχους που θέλουμε να υλοποιήσουμε στο μέλλον, πολύ φοβούμε ότι δεν μπορούμε να μιλούμε για αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της ΚΑΠ, αν δεν έχουμε προηγουμένως προσυμφωνήσει τους στόχους. Γιατί η αποτελεσματικότητα αφορά τους στόχους τι θέλουμε να επιδιώξουμε, τι επιδιώκουμε, τι θέλουμε να επιτύχουμε, να πραγματοποιήσουμε με την ΚΑΠ. Θέλουμε καλύτερη παραγωγικότητα, αυτό είναι ο στόχος μας. Θέλουμε καλύτερη κερδοφορία της γεωργίας, είναι αυτός ο στόχος. Θέλουμε καλύτερη διαβίωση, καλύτερο βιωτικό επίπεδο των γεωργών. Θέλουμε καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος. Ποιοι είναι οι βασικοί μας στόχοι για την κοινή γεωργική πολιτική και πώς συνδέονται μεταξύ τους. Αν ε, οι νομοθέτες δεν έχουν στο μυαλό τους με αυτά τα θέματα, τους στόχους, θα είναι δύσκολο να κρίνουμε με κάποιο γνώμονα την κοινή πολιτική. Αυτό είναι το πίσω ζήτημα λοιπόν, οι στόχοι. Το πρώτο και πιο σημαντικό. Δεύτερο σημαντικό ζήτημα. Και θα τα πω στα γαλλικά αυτή τη φορά. Γιατί η ερώτηση έγινε στα γαλλικά. Για το ιστορικό μοντέλο, για τα ιστορικά σημεία αναφοράς. Όλοι γνωρίζουμε ότι η κοινή γεωργική πολιτική είναι η παλαιότερη κοινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρώτη κοινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γνωρίζουμε ότι από το 2003 ανακύπτει το πρόβλημα των ιστορικών σημείων αναφοράς, του ιστορικού μοντέλου για τις δημόσιες επιδοτήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ε, αναφέρονται στο 2003 και περιλαμβάνονται και στη μεταρρύθμιση του 2013 και θα φανούν και στα αποτελέσματα του 2019 και του 2020 αυτές οι ιστορικές αναφορές. Γνωρίζουμε επίσης ότι τα κράτη-μέλη υιοθέτησαν διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλογα με τις δυνατότητες που τους έδινε η Ευρωπαϊκή Ενωσιακή Νομοθεσία. Οπότε το ζήτημα που θα ανακύψει στο μέλλον είναι θα συνεχίσουμε στο μέλλον να διαχειριζόμαστε τα ιστορικά προβλήματα του παρελθόντος. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να προβληματίσει τον Ευρωπαίο νομοθέτη. Περνάω ξανά στα αγγλικά. Τρίτο ζήτημα σημαντικό που ανακύπτει από το δικό σας προβληματισμό. Το θέμα της ανταγωνιστικότητας. Τι επιδιώκει πραγματικά ο νομοθέτης για το μέλλον και την ανταγωνιστικότητα. Ένας εξωτερικός παρατηρητής, σαν και εμένα, ένας δημόσιος ελεγκτής, όπως και εγώ, βλέπει με σαφήνεια τι επιδιώκει με την εσωτερική σύγκληση ο νομοθέτης. Επίσης, είναι και φαίνεται προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να υλοποιήσουμε αυτή την εσωτερική σύγκληση. Αλλά δεν ξέρω τι θέλει στο μέλλον ο νομοθέτης ως προς την εξωτερική σύγκληση. Και αυτό είναι μια και δική μου απορία. Λυπάμαι γιατί σας απαντώ και εγώ με ερωτήσεις, αντί να σας δίνω απαντήσεις στις ειδικές σας ερωτήσεις. Αλλά σας θέτω και εγώ ερωτήσεις, γιατί εσείς είστε ε, οι νομοθέτες. Οπότε εσείς θα πρέπει να βρείτε τις απαντήσεις, γιατί οι απαντήσεις αυτές έχουν πολιτικό χαρακτήρα. Οπότε το θέμα της εσωτερικής σύγκλησης είναι πολύ σημαντικό, της σύγκλησης. Τέταρτο σημαντικό ζήτημα, το θέμα των αποσυνδεδεμένων ενισχύσεων. Κάποιος ευρωβουλευτής με ρώτησε, θα συνεχίσουμε με τις αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις ή θα πρέπει να περάσουμε σε ένα μοντέλο συνδεδεμένων ενισχύσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διεθνείς υποχρεώσεις, διεθνείς ανηλυμένες υποχρεώσεις. Οπότε, όπως είπε κάποιος άλλος ευρωβουλευτής, πριν από λίγο, θα πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι η Ευρωπαϊκή Γεωργία πρέπει να είναι ανταγωνιστική παγκοσμίω, γιατί στο παγκόσμιο προσκήνιο δραστηριοποιείται. Και σε αυτό το παγκόσμιο επίπεδο έχουμε αναλάβει κάποιες υποχρεώσεις και θα πρέπει να τις στηρίσουμε. Πέμπτο μείζον ζήτημα αφορά τη στόχευση. Και είναι συναφές και με το ζήτημα της αποτελεσματικότητας. Τα χρήματα μας πιάνουν τόπο. Δηλαδή, επιφέρουν αποτελέσματα, αποφέρουν καρπούς. Και στην συγκεκριμένη ειδική έκθεση και σε άλλες ειδικές εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου φαίνεται ότι έχουμε αμφιβολίες ως προς την αποτελεσματικότητα, ως προς το αν πιάνουν τόπο τα κονδύλια της ΚΑΠ. Άλλο θέμα αφορά την απλοποίηση, την απλούστευση. Αυτό που βλέπουμε στην ειδική μας έκθεση είναι ότι όταν τα κράτη-μέλη ανέλαβαν κάποιες αρμοδιότητες για να κάνουν επιλογές και κάποια διακριτική ευχέρεια για να αναπτύσσουν πλαίσια, σε μερικές περιπτώσεις τα κράτη-μέρη χρησιμοποίησαν αυτές τις εξουσίες όχι για να απλουστεύσουν την ΚΑΠ, αλλά για να την περιπλέξουν. Οπότε το αφήγημα ότι οι κανόνες των Βρυξελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι που περιπλέκουν τα πράγματα, ε, δεν ισχύει. Τα κράτη-μέλη πολλές φορές ευθύνονται για την ε, περιπλοκή της ΚΑΠ, για την αύξηση της περιπλοκότητας. Επίσης, το θέμα της ισότητας. Αυτό φορά εν μέρη και την εξωτερική σύγκληση και την αποτελεσματικότητα. Και γαλλικά και πάλι το θέμα του γενικού, του σφαιρικού οράματος το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ήδη έχει εκπονήσει πολύ άριθμες εκθέσεις για την κοινή γεωργική πολιτική. Η συγκεκριμένη δική έκθεση για το καθεστώς βασικών ενισχύσεων αφορά ακριβώς αυτό το θέμα, αλλά υπάρχουν πολλές άλλες εκθέσεις που αφορούν άλλα θέματα. Την οικολογικοποίηση, Φερρυπίν, την αγροτική ανάπτυξη, τους νεαρούς αγρότες, έχουμε πολλές εκθέσεις, δεκάδες εκθέσεις για τους νεαρούς αγρότες. Πάντως, αυτό που κάναμε για το γενικό όραμα είναι να σας να συντάξουμε το έγγραφο που θα σας παρουσιάσω σε λίγο, στο σημείο 5 αντιδρώντας στην ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας. Οπότε αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε και έχουμε λίγο χρόνο, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο για να προσθέσει κάποιες λεπτομέρειες στα θέματα αυτά. Αν μου επιτρέπετε φυσικά κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κάποια ερωτήματα τεχνικού χαρακτήρα και θα ήθελα, και θα ήθελα να εξηγήσω πολύ σύντομα τι διαπιστώσαμε κατά τον έλεγχο για τις ε, μόνιμες χορτολιβαδικές ε, εκτάσεις που δεν στοχεύσε ιδιαίτερο ελεγχός μας γιατί εμείς κοιτάξαμε το συνολικό υπολογισμό ε, των εκτάσεων που μπορούσαν να είναι δικαιούχοι. Σημειώθηκε πάντως από την έκθεση αλλά και σε σχέση με τους χαλακτών παραγωγούς που αναφέρθηκαν νωρίτερα και που αντιμετώπισαν την τελευταία κρίση το εξής. ότι υπήρχε θέμα με τι επαγγελματικέ εκτάσει. Επίση, σε σύγκληση έγινε νομίζω διεξοδική αναφορά. Ένα άλλο σημαντικό θέμα αφορά την αναγκαιότητα να καλύπτονται οι προϋποθέσεις για τους δικαιούχους των ενισχύσεων και ιδιαίτερα όσον αφορά για την, καταπο, την καταποκοπή ενίσχυση. Το έχουμε συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία επιμένει ότι απαιτείται για να, και για όρους συμμόρφωσης ε, με τη Συμφωνία ΠΟΕ. Στην απλούστευση, η απλούστευση αφενός και η στόχευση αφετέρου. Έχουμε κάποια παραδείγματα στην έκθεση για τη Γαλλία, επί παραδείγματι και την Ισπανία, όπου βλέπουμε ότι κάποιες επιλογές των κρατών οδήγησαν σε αύξηση του περιπλοκού των διαδικασιών για τον Γεωργό και του τρόπου με τον οποίο ο Γεωργός αντιλαμβάνεται το σύστημα. Η Γαλλία είναι ένα ενδιαφέρον παράδειγμα. για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να περιπλακεί ένα σύστημα με την εισαγωγή διαφόρων κανόνων ε, παραδείγματι χαρακτηριστικά τοπίου που μπαίνουν στην οικολογικοποίηση σε έναν βαθμό μπορεί να περιπλέξουν πολύ το, την εφαρμογή του συστήματος. Και από την άλλη είδαμε και συστήματα που απλοποιούν περισσότερο την κατάσταση στα κράτη-μέλη χωρίς να είναι λιγότερο αποτελεσματικά. Η αποσύνδεση των ενισχύσεων για την ε, υποστήριξη των αγορών και μηχανισμών αγοράς. Στην ε, αποσυνδεδεμένη ενίσχυση ε, εισοδήματος πηγαίνει τώρα το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού και με τις αναδιανομητικές πληρωμές και με την οικολογική οικολογικοποίηση κτλ. Βεβαίω θα πρέπει η Επιτροπή να επιλέξει ποιος είναι ο καλύτερος, καταλληλότερος, πιο αποτελεσματικός τρόπος να στηριχθεί το εισόδημα των γεωργών συνδυάζοντα αυτά τα... Να, να υποστηριχθεί το εισόδημα των γεωργών. Νομίζω δεν ξέχασα τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και ελπίζω στις πολυάριθμες ερωτήσεις σας να δώσαμε κάποιες απαντήσεις. Φυσικά, αν δεν είστε ικανοποιημένοι, μέσα στη διάθεσή σας για περισσότερες απαντήσεις. Και σε, άλλα, και σε διάφορα κέντρα συζητήσεων πρέπει να πω. Ευχαριστώ λοιπόν για τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις των ε, βουλευτών αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστούμε κύριε Φιγκερέντο. Νομίζω ότι αυτό το θέμα το εξαντλήσαμε. Χωρίς καν να χρειαστεί να περιορίσουμε το χρόνο αγόρευσης. Είχαμε την πολυτέλεια του χρόνου σήμερα. Σας ευχαριστούμε και πάλι κύριε Φιγκερέντο. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το σημείο 5 δεύτερο ουσιαστικό θέμα της σημερινής διάταξης που αφορά και πάλι μια παρουσίαση του κυρίου Φιγκερέντο από το Ελεκτικό Συνέδριο. Θα μας παρουσιάσει τη σκέψη του για το μέλλον της κοινή γεωρικής πολιτικής μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Νοεμβρίου 2017 για το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας. με μεγάλη χαρά θα ξανακούσουμε τον κύριο Φιγκερέντο. Χωρίς άλλη χρονοτριβή, θα ξαναδώσω και πάλι το λόγο στον καλεσμένο μας. Thank you, Mr. Σας ευχαριστώ και πάλι κύριε Πρόεδρε που μας δίνεται τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε στα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας ένα έγγραφο το οποίο προετοιμάσαμε σε μικρόχρονικό διάστημα ερχόμενη σε ε, απάντηση της ανακοίνωσης της Επιτροπής για το μέλλον της ΚΑΠΑ. Έχω και πάλι ετοιμάσει μια παρουσίαση για τη διευκόλυνση της συζήτησής μας και το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι αυτό το υπόμνημα, αυτή, αυτό, το έγγραφο έρχεται σε απάντηση της, στην ανακοίνωση της Επιτροπής για το Μέλλον της, ε, των Τροφίμων και της Γεωργίας. Δεν είναι ελεγκτική έκθεση, είναι μια ανασκόπηση προηγούμενων εκθέσεων και εκδόσεων του ελεγκτικού συνεδρίου, καθώς επίσης και άλλων πληροφοριών που είναι δημοσίως διαθέσιμες. Δηλαδή, ε, συνοψίζουμε ε, αυτά που είχαν δημοσιοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Σε αυτό το έγγραφο, λοιπόν, εστιάζουμε σε τάσεις και δεδομένα, τα οποία έχουν κρίσιμη σημασία για την γεωργία και για τις γεωργικές περιοχές, την περιφέρεια, τα ευρήματά μας όσον αφορά την τρέχουσα κοινή αγροτική πολιτική επί τη βάση των προηγούμενων εκθέσεων του Ελεκτικού Συνεδρίου και τρίτον σε κριτήρια και προκλήσεις που θεωρούμε ότι θα πρέπει να λάβει υπόψη τη χάραξη της νέας ΚΑΠ. Βεβαίως, δεν είναι ο ρόλος του Ελεκτικού συνεδρίου να κάνει προτάσεις πολιτικής. Αλλά ε, αξιοποιούμε την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει από τους ελέγχους μας, από τα ευρήματά τους, για να επισημάνουμε ορισμένα στοιχεία. Όσον αφορά τώρα τις τάσεις και τα δεδομένα που έχουν ιδιαίτερη σημασία. Το πρώτο που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι την τελευταία δεκαετία οι δαπάνες για την ΚΑΠ έχουν παραμείνει σταθερές κατά μέσον όρο 54 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αυτό ε, το ποσό έχει παραμείνει σταθερό στο, οι δημόσιε δαπάνε στον τομέα αυτών έχουν παραμείνει σταθερέ και το βλέπετε αυτό και στην γραφική παράσταση που επιπροσθέτω δείχνει και την κατανομή στου επιμέρου τομεί. Βλέπετε ξεκάθαρα ότι υπάρχει σταθερότητα. Επομένω, μία πρόταση που είναι και το πρώτο σημαντικό στοιχείο της, ε, του εγγράφου μα, Μία πρόταση για αύξηση των δαπανών κατά 350 δισεκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να δικαιολογηθεί πλήρως και προσεκτικά. Θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δαπανά του τα κονδύλια της ΚΑΠ στο μέλλον ε, σε μέτρα τα οποία να έχουν βασιστεί σε στατιστικά στοιχεία και σε επιστημονικά στοιχεία που να μας αποδεικνύουν ότι τα μέτρα αυτά θα έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα που θα μας αποδεικνύουν ότι θα, είναι, θα υπάρχει αποτελεσματικότητα στην οποία αναφέρθηκα και προηγουμένως άλλα σημαντικά στατιστικά στοιχεία και, και τάσεις. Δείτε στο γραφική παράσταση αυτή. Είναι στοιχεία τα οποία έχουμε πάρει από την ανακοίνωση της Επιτροπής και είναι στοιχεία τα οποία αναφέρονται στο εισόδημα των αγροτών. Όμω, καλύπτονται και συμπεριλαμβάνονται όλε οι εκμεταλλεύσει, ακόμα και εκείνε οι οποίε είναι πολύ μικρέ και δεν αποφελούνται ω εκ τούτου από την ΚΑΠ και δεν γίνεται καμία διάκριση μεταξύ του μεγέθου, του οικονομικού τη εκμετάλλευση. Η γραφική παράσταση αυτή που έρχεται λοιπόν από την Επιτροπή μα ε, δείχνει ε, και το χρησιμοποιεί αυτό το επιχείρημα η Επιτροπή για να μα πει ότι το εισόδημα το αγροτικό υπολείπεται ακόμα του μέσου εισοδήματο, στη μισθωτή εργασία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλε τι οικονομίε τη. Όμω έχουν συμπεριληφθεί όλε οι αγροτικέ εκμεταλλεύσει, ακόμα και εκείνες οι οποίε είναι πολύ μικρέ και ω εκ τούτου δεν ε, εποφελούνται από την ε, ΚΑΠ. επίση δεν συνυπολογίζονται άλλα εισοδήματα πέραν των γεωργικών που ίσω να έχουν ε, οι αγρότες. Το επισημαίνουμε λοιπόν αυτό ως ε, έναν περιορισμό των συμπερασμάτων που μπορεί να εξάγει κανείς από αυτή τη γραφική παράσταση. Κάτι ακόμα, μια ακόμα γραφική παράσταση που μας δείχνει τις τάσεις. Βλέπουμε με την ε, σκούρα μπλε γραμμή ότι έχει μειωθεί ο αριθμός των αγροτών σε σχέση με το παρελθόν με την γαλάζια γραμμή, την ενδιάμεσου της απόχρωσης, γαλάζια γραμμή, βλέπετε ε, το ποσοστό της απασχόλησης στον γεωργικό τομέα. Συγγνώμη, αυτή ήταν η ανοιχτή γαλάζια γραμμή. Και στη μεσαία γραμμή βλέπετε ε, ποιο είναι το ε, οικονομικό αποτέλεσμα αυτών των εκμεταλλεύσεων. Τι μπορούμε να συμπεράνουμε από αυτή τη γραφική παράσταση. Βλέπουμε ότι λιγότερες και μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις δημιουργούν ένα σταθερό οικονομικό αποτέλεσμα, το οποίο σημαίνει ότι το κατακεφαλήν εισόδημα εκείνων που απασχολούνται στον τομέα της γεωργίας αυξάνεται. Αυτό είναι μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με το τι συνέβαινε στο παρελθόν. Άλλες σημαντικές ε, τάσεις ε, και στοιχεία στατιστικά μας δείχνουν ότι πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει καθαρός εξαγωγέας ε, τροφίμων, συνεχίζει όμως να είναι ε, καθαρός εξαγωγές των ε, μη επεξεργασμένων αγροτικών προϊόντων. Συνεχίζει να εισάγει τέτοια προϊόντα. Επίσης διαπιστώνουμε ότι ο μέσος όρος ηλικίας των αγροτών αγροτών, των, των διαχειριστών μάλλον των αγροτικών εκμεταλλεύσεων έχει αυξηθεί και ακολουθεί τις γενικότερες δημογραφικές τάσεις. Ωστόσο, τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας για τη συνολική έκταση που χρησιμοποιείται για γεωργική παραγωγή ε, δεν είναι συνεκτικά, δεν μας δείχνουν μια καθαρή εικόνα, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εάν αυξάνεται αυτή η έκταση ή αν μειώνεται συνολικά. Εάν κοιτάξουμε στο στατιστικό, στα στατιστικά στοιχεία που αφορούν το, ποσότητες της ε, ίσω φαίνεται να υπάρχει μια μείωση τη τάξη του 4%. Αλλά δεν είναι ξεκάθαρα τα στοιχεία αυτά. Επίσης διαπιστώνουμε ότι η πρόοδο όσον αφορά τα μέτρα για την καταπολέμηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων δεν είναι ικανοποιητική. Και όπω είπα προηγουμένω, έχει μειωθεί η ψαλίδα ε, ανάμεσα στις, ε, στην αγροτική περιφέρεια ε, και στι άλλε περιφέρειε, στις αστικέ. οι μελλοντικές προτάσεις για την εξέλιξη της κοινή αγροτικής πολιτικής. Κατά την άποψή μας θα έπρεπε να ακολουθήσουν μια δομή ε, λογική η οποία θα, σας βοηθήσει, θα βοηθήσει και το δημόσιο διάλογο αλλά και εσάς το συνομοθέτη. Και σας παρουσιάζω το μοντέλο που εμείς προτείνουμε. Πρέπει να ξεκινήσουμε από έναν εντοπισμό των αναγκών που έχουμε στον τομέα της γεωργίας. Μετά να πάμε στους στόχους που θέλουμε να καθορίσουμε, τους στόχους μας για το μέλλον. Να δούμε μετά τι παρεμβάσεις θα είναι ε, ε, επιβεβλημένες, με ποιες διαδικασίες και σε τι αποτελέσματα θα οδηγήσουν αυτές. Τι αποτελέσματα θα έχουν οι παρεμβάσεις μας στο μέλλον. Ε, αυτό το μοντέλο σκέψης μπορούμε να αξιολογήσουμε την τρέχουσα ΚΑΠ αλλά και τις όποιες προτάσεις έρθουν για το μέλλον της ΚΑΠ. Οι στόχοι της ΚΑΠ θα πρέπει να ανταποκρίνονται τους, στο μακροπρόθεσμο όραμα και στους, ε, στις βασικές ανάγκες που έχουν εντοπιστεί και μετά να μεταφράζονται σε ποσοτικοποιημένους στόχους αντικτύπου και αποτελεσματών. Επίσης θα χρειαστούμε ένα μηχανισμό για την ε, τακτική επαναξιολόγηση της πολιτικής αυτής που λειτουργεί ουσιαστικά και επίσης ένα πλήρες πλαίσιο για τη λογοδοσία όσων συμμετέχουν στην εφαρμογή της πολιτικής. Όσον αφορά τις ανάγκες. Λέμε ότι δεν έχουμε στα χέρια μας επαρκή στοιχεία έτσι ώστε να μπορούμε να εντοπίσουμε Ποιε είναι συγκεκριμένε ανάγκε και να μπορούμε να δικαιολογήσουμε όλη τη δαπάνη που γίνεται με τη σημερινή ΚΑΠ. Θα πρέπει κατά την άποψή μα επίση να διευκρινιστεί περισσότερο η έννοια τη προστεθέμενη αξία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίση, η ΚΑΠ θα πρέπει να μπορεί να ανταποκρίνεται καλύτερα στι πιο μακροπρόθεσμες εξελίξει και τάσει. Σε αφορά τώρα του στόχου. Πιστεύουμε ότι οι τρέχοντες στόχοι της ΚΑΠ δεν είναι αρκετά ξεκάθαροι και επίσης οι πολιτικοί, πολιτικοί στόχοι της κοινή αγροτικής πολιτικής θα πρέπει να είναι συνεκτικοί, να ταιριάζουν με, με, με, με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Άνωσης σε άλλους τομείς πολιτικής. Επίσης, αυτή τη στιγμή ε, οι παρεμβάσεις που γίνονται δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι δικαιολογούνται πάντοτε ε, και δεν αποδεικνύεται πάντα η προστεθέμενη εξαίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τώρα τις διαδικασίες. Για να μπορούμε να σχεδιάζουμε μέτρα στο, στο πλαίσιο της ΚΑΠ χρειαζόμαστε καλύτερες πληροφορίες και πιο γρήγορα. Πρέπει να βελτιώσουμε επίσης τη συνεκτικότητα ανάμεσα στην ΚΑΠ και τις άλλες πολιτικές της Ένωσης, καθώς επίσης και ανάμεσα στα διάφορα μέτρα της ΚΑΠ μεταξύ τους. Η πολιτική θα πρέπει να απλοποιηθεί, χωρίς όμως αυτό να λειτουργήσει εις βάρος της αποτελεσματικότητας. Και επίσης ε, πιστεύουμε ότι η υιοθέτηση και η εφαρμογή μιας νέας ΚΑΠ, μιας μεταρρυθμισμένης ΚΑΠ, χρειάζεται χρόνο για να αποδώσει. Σε σχέση με τους εξωτερικούς παράγοντες, καθώς επίσης και με τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Θεωρούμε ως ελεκτικό συνέδριο ότι το σημερινό σύστημα δικτών που έχουμε δεν είναι επαρκές και δεν μας επιτρέπει να αξιολογούμε την πολιτική μας και τις επιδόσεις μας. Δεν χρειάζεται να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη σχέση εντοπίσει ανάμεσα στη δαπάνη φαινός και στο αποτέλεσμα αφετέρου. Τέλος, πρέπει να ενισχύσουμε την λογοδοσία στον τομέα της κοινής αγροτικής πολιτικής. Αυτά που σας παρουσίασα έως τώρα είναι τα συμπεράσματά μας, τα... οι απόψεις μας για τη σημερινή ΚΑΠ. Έχουμε επίσης και κάποιες, ε, καμιά παρόμοια ανάλυση όσον αφορά το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής κοιτώντας στα στάδια που σας είπα, τους εξωτερικούς παράγοντες, ε, τις παρεμβάσεις που επιθυμούμε να κάνουμε, τις ανάγκες που πρέπει να καλύψουμε, τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα που επιδιώκουμε. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες, όμως ήθελα να επισημάνω ότι με αυτά τα κριτήρια ε, θα αξιολογήσει το ελεκτικό συνέδριο στο μέλλον τις προτάσεις για την ΚΑΠ. Και ίσως, κατά την άποψή μας, τα κριτήρια αυτά θα είναι χρήσιμα και για τους συνομοθέτη όταν εσείς λάβετε αυτές τις προτάσεις και τις αξιολογήσετε τη δική σας την πλευρά σας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Φιγκερέντο, κύριος Ντες. Αυτή τη φορά ε, να είμαστε πιο σύντομοι. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ και για αυτή την έκθεση. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπα και νωρίτερα, τα 54 δισεκατομμύρια ευρώ που δίνουμε για την Ευρωπαϊκή Γεωργία δεν κατανέμονται δίκαια, το είπαν και οι συνάδελφοι, θα τους δώσω δίκαιο. Ωστόσο αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι η Γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχεί σε 41 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και βέβαια προσφέρει σε 500 εκατομμύρια πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης καθημερινά υγιή τρόφιμα και καθαρά τρόφιμα. Εγώ 40 χρόνια ασχολούμαι με τη γεωργική πολιτική. 40 χρόνια μελετώ τα θέματα αυτά. Βλέπω λοιπόν ότι δεν ε, ε, αυξάνεται ο χρόνος εργασίας ο ημερήσιος στην ε, γεωργία όπως σε άλλους τομείς απασχόληση ενδεχομένως. Εδώ και δεκαετίες βλέπουμε να μειώνεται μάλιστα ο χρόνος, οι ανθρωπόρες δηλαδή, γιατί είναι πολλοί οι γεωργοί που εγκαταλείπουν το επάγγελμα. Ε, γιατί, διότι τους έχουμε κατακλείσει με υπερβολικά πολλές απαιτήσει και κανονισμούς πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν πλέον να διαχειριστούν τις επιχειρήσεις τους και εγκαταλείπουν τη γεωργική δραστηριότητα. Ε, έχουν να υποστούν ε, τις ε, τους περιορισμούς των διαφορών διατάξεων για την προστασία των ζώων και άλλους κανονισμούς. Πολλοί είναι αυτοί λοιπόν οι οποίοι κλείνουν τις ε, τους εκμεταλλεύσεις που εγκαταλείπουν την γαλακτοπαραγωγή. Λίγοι είναι οι νέοι οι οποίοι δεν είναι οι οποίοι πλέον θα ήταν διατεθειμένοι και αυτό οφείλεται και στην οικονομική κατάσταση να αναλάβουν το επάγγελμα του γεωργού. Και έχει τύχει να συναντήσω μια οικογένεια όπου ο πατέρας ήταν γεωργός, ο νέος, ο νεαρός γιος είχε μάθει το επάγγελμα, αλλά αποφάσισε μετά, όπως μου είπε ο πατέρας, να μην ε, το ασκήσει γιατί δεν μπορούσε να επιβιώσει από αυτό. Θέλω και για να είμαι σύντομος να αναφερθώ σε μια μελέτη της δεκαετίας του 90 στην Γεωργία, η οποία αναφερόταν, η οποία εξέθεται τις, όλα τα ωφέλη της γεωργίας και όχι μόνο καθαρά στην γεωργική παραγωγή. Αυτή νομίζω την έκθεση πρέπει να έχει υπόψη το λεκτικό συνέδριο. Ευχαριστώ. Αγαπητέ Άλμπερτ Ντες, δεν ε, νομίζω ότι εξυπηρετήσε τίποτα να λέμε ότι είναι λίγα τα χρήματα. Είναι ένα ποσοστό του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφου από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που ορίζουν έτσι τις προτεραιότητες και την ε, αναλογία της χρηματοδότηση από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό που πηγαίνει στην ε, γεωργική ε, πολιτική. Για την ε, μελέτη που ανέφερε τη βαβαρία είναι του 90 όμω, έχουν περάσει εδώ μεταξύ κοντά 30 χρόνια. Για το ελεγκτικό συνέδριο. Πολύ σωστά επισημαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα στην αξιολόγηση των στοιχείων, αλλά δεν συμφωνώ ότι δεν έχουμε αρκετά στοιχεία. Ξέρουμε ότι μειώνει το αριθμό των γεωργών. Ξέρουμε ότι είναι όλο και τώρα οι μεγάλε εκμεταλλεύσει. Ε, γιατί λοιπόν δεν προχωρείτε και στο επόμενο βήμα και να πείτε ότι οι στόχοι δεν υλοποιούνται όπως πρέπει. Και θα ξαναναφέρω βέβαια το περιβάλλον. Αυτή η κοινή γεωργική πολιτική δεν μπορεί να εξαντλείται στο ε, να είναι μόνο ένα σύστημα ή ένα μέσον κάλυψης εισοδηματικών αναγκών. Εάν δεν υπηρετήσουμε όλους τους στόχους και βέβαια δεν εξασφαλίσουμε και ένα αξιοπρεπές εισόδημα για τον παραγωγό, δεν έχει κανένα νόημα αυτή η πολιτική. Πρέπει να οριστούν στόχοι λοιπόν. Και σας καλώ με θάρρος να πείτε ξεκάθαρο ότι το δημόσιο χρήμα είναι και αυτό το οποίο θα υπηρετήσει τα δημόσια αγαθά. Και σε αυτό θα πρέπει να στοχεύει. Δεν μπορούμε να προσποιούμε ότι αυτή η γεωργική πολιτική, τουλάχιστον έτσι είναι αυτό, είναι μόνο ένα μέσον αναδιανομής χρήματος για τη διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα και άρα ο γεωργικός τομέας καλύπτεται σε σχέση με τα έσοδα τα οποία χάνει γιατί δεν είναι αρκετά ανταγωνιστικό στις διεθνείς αγορές. Γιατί και 60 και 80 δισεκατομμύρια να δώσω πάλι δεν θα φτάσουν. Βεβαίω πρέπει να οριστούν προτεραιότητε. και αυτό είναι πολιτικό καθήκον το οποίο βεβαίως δεν μπορεί να υλοποιήσει το ελεκτικό συνέδριο ως εκ του, αλλά πολιτικά, πολιτικούς στόχους και πολιτικές επιλογές πρέπει να κάνουμε εμείς για να υπηρετήσουμε το φορολογούμενο με τα κριτήρια που θα οριστούν. Και αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Γιλέρα. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε καλύτερα πώς βλέπετε αυτή τη θετική κατέθεση των ε, στρατηγικών σχεδίων για την ε, μελλοντική πολιτική. Εμένα με προβληματίζει η στρέβλωση της αγοράς και από περιβαλλοντική άποψη και από άποψη προϊόντων. Νομίζω ότι είναι πολύ πρόημη αυτή η θετική εικόνα που δίνεται για τα στρατικά, στρατηγικά σχέδια. Επίσης, στα κράτη-μέλη υπάρχουν διαφορετικές αρμοδιότητες. Έχουμε και τοπική αυτοδιοίκηση πολλές φορές ε, με σημαντικές αρμοδιότητες. Οπότε το, το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο δεν έχει την ισχύ συντάγματο σε περίπτωση που υπάρχουν και περιφερειακές ή ορικές αρμοδιότητες. Θέλω περισσότερα στοιχεία για τη δήλωση που μας κάνατε. Επίσης, μιλήστε για αναδιανεμητικές ε, ενισχύσεις ή πληρωμέ είπατε ότι δεν αποφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Εξετάστε και την πιθανότητα να περιορίσετε τις βασικές ενισχύσεις με ένα νότατο όριο και μετά να κάνουμε την αναδιανομή. Γιατί στη δική σας ανάλυση θεωρείτε ότι οι αναδημητικές πληρωμές δεν είχαν τα ε, αναμενόμενα αποτελέσματα. Το κάπινγκ, η υποβολή έχει, έχει πολιτικό χαρακτήρα, αλλά ποιες θα είναι οι συνέπειες ε, των αναποτελεσματικών αυτών αναδιανεμητικών ε, πληρωμών. Μήπως ε, τα αποτελέσματα της αναδιανομής δεν ήταν σωστά προσδιορισμένα. Εσείς τι ανάλυση κάνατε, ο κύριος Κάρθη. Ευχαριστώ και ευχαριστώ το Ελεκτικό Συνέδριο για την παρουσίαση αυτής της έκθεσης που είναι, έχει ιδιαίτερα πολιτικό χαρακτήρα. Φαντάζομαι θα συμφωνούν οι συνάδελφοι. Ε, η έκθεση μιλάει για καλύτερη στόχευση, για στόχους που θα στηρίζονται σε συγκεκριμένα στοιχεία και αποδείξεις. Συμφωνώ. Επίσης, θε... πολλές φορές ε, ζητούμε περικοπές σε περίπτωση που δεν προσφέρεται προστιθέμενη αξία ευρωπαϊκή. Πολύ φοβάμαι όμως ότι είναι διαφορετική αντίληψη για το τι εστί θεμενή αξία. Για παράδειγμα, είπαμε ότι η κοινή γεωργική πολιτική θέλει να εξασφαλίσει αξιοπρεπέ βιωτικό επίπεδο της, ε, του γεωργικού πληθυσμού και η ενίσχυση του κοινωνικο-οικονομικού ιστού τη υπαίθρου. Αυτό όμω δεν συνάδει με αυτό που εσεί καθορίζετε ω προ τη θεμενή αξία και πώ τον υπολογίζετε. Επίσης, αναφέρεται ότι έχουμε σήμερα 22% λιγότερους γεωργούς από ότι το 2007. Φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη μαζική αποχώρηση, έξοδος από τις, από τις γεωργικές κοινότητες, κυρίως από εγκατάλειψη των μικρομεσαίων γεωργών. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Μήπως θα μπορούσατε να μας δώσετε μια πιο συγκεκριμένη απάντηση για το τι εσείς θεωρείτε ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Ιδιαίτερα όταν θέλετε αυτό να συμπεριληφθεί στα μέτρα χρηματοδότηση αυτό το κριτήριο. Ε, υπάρχουν πολλές σημείες για τον ε, προϋπολογισμό που θα εδράζεται στις επιδόσεις και συνδέεται ε, τους πόρους με την υλοποίηση των αποτελεσμάτων. Αυτό όμω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δήλωσε ως ε, ασύμβατο προ προς τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Πώς είναι δυνατόν να μειώσουμε την ανασφάλεια, την αβεβαιότητα των γεωργών που κάθε χρόνο θα φοβούνται ότι θα κοπούν οι πληρωμές αν δεν υλοποιηθούν κάποιοι στόχοι. Έτσι θα αυξηθεί η έξοδος από τη γεωρική δραστηριότητα, κάτι που θέλουμε να αποτρέψουμε κανονικά. Τέλος, κάτι που φαίνεται ως σκεπτικισμός στην έκθεση ότι τα γεωργικά εισοδήματα είναι χαμηλότερα από το μέσο όρο των εισοδημάτων άλλων οικονομικών κλάδων. Δεν ξέρω τι σημαίνει σε άλλε χώρε. Πάντω στην Ιρλανδία το ετήσιο ε, γεωργικό εισόδημα είναι 20.000, ενώ το βιομηχανικό είναι 37.000 για του απασχολούμενου στη βιομηχανία. Βέβαια, μερικοί λένε ότι μερικοί γεωργοί κρύβουν ε, κάτω τα στρώματά του ε, τι οικονομίε του. Αλλά φαντάζομαι δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι κάτι τέτοιο ισχύει, ότι έχουν κρυφά εισοδήματα. Επίσης, ε, τονίζεται ότι πολλοί γεωργοί έχουν και μη γεωργική δραστηριότητα. Ε, υπό 30.000 είναι αυτοί που έχουν εξωγεωργική δραστηριότητα και αμοιβή. Βέβαια, οι περισσότεροι γεωργοί θέλουν να είναι γεωργοί και να έχουν αποκλειστικά γεωργικά εισοδήματα. Αλλά μόνο τα γεωργικά εισοδήματα δεν του επιτρέπουν το βιοπορισμό και την επιβίωση. Γι' αυτό μερικέ παρεστρέφονται σε έξω γεωργικέ δραστηριότητε. Μερικέ φορές μάλιστα το χαμηλό κόστος παραγωγής, ε, η πόλη του κόστος κάτω του κόστος παραγωγής του γονατίζει. Είχαμε πολλές συζητήσεις ε, στην Επιτροπή Γεωργία ω προς την ανάγκη να ε, ενημερώσουμε, να καταρτήσουμε, να διαπαιδαγωγήσουμε τον καταναλωτή για τη σημασία και τις αξίες της ΚΑΠ. Ίσως θα πρέπει να επεκτείνουμε την ε, διαπαιδαγώγηση και στα άλλα κοινοτικά θεσμικά όργανα και στο ελεκτικό συνέδριο, γιατί υπάρχει μεγάλο κενό μεταξύ της θεωρίας της έκθεσης και της πραγματικότητας στην Ήπεθρο και στη Γεωργία. Ευχαριστώ κύριε Σουλαζό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί εκπρόσωποι του ελεκτικού συνεδρίου, εγώ θα ήθελα να σταθώ ακριβώς στο ε, στοιχείο της μείωσης του αριθμού του, των εκμεταλλεύσεων και επίσης ότι έχουν αυξηθεί, το έχει αυξηθεί κατά 28% το μέγεθός τους, το οποίο είναι, ε, έχει ως ε, αποτέλεσμα να ε, μειώνεται η θέσεις εργασίας. Λέτε ότι το οικονομικό αποτέλεσμα έχει παραμείνει σταθερό και ε, ως εκ τούτου λέτε ότι το μέσο εισόδημα του γεωργικού αυξάνεται. Και θα ήθελα να μου πείτε για ποιες ε, χώρες μιλάτε. Είναι ορισμένες οι οποίες είναι ιδιαίτερα προνομιούχες, αλλά η δικιά μας εμπειρία είναι ότι στην πραγματικότητα όπως βλέπουμε στη Γαλλία, οι επιδοτήσεις μειώνονται, τα εισοδήματα τα αγροτικά μειώνονται. Ίσως ε, βέβαια να μιλάτε για ορισμένες άλλες χώρες οι οποίες να επιθυμούν να γίνουν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μας πείτε. έχουμε μία τάση να πηγαίνουμε περισσότερο προς την βιομηχανοποιημένη, την, ε, την τυποποιημένη γεωργία και δεν μιλούμε για τα βιολογικά προϊόντα. Επομένως, κατά την άποψή μου δεν έχετε υπόψη σας το πραγματικό συμφέρον και την πραγματικότητα και την καθημερινότητα των αγροτών σε χώρες όπως τη Γαλλία παρά μόνο στις στατιστικές σας. Κύριος Κάστρο, εγώ θα ήθελα, Πρόεδρε, ευχαριστώντα βέβαια τους εκπροσώπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις τοποθετήσεις τους, να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Ε, τους στόχους ε, τους ορίζει η συνθήκη, αγαπητοί συνάδελφοι. Προστασία του Γεωργού. Και αυτό ορίζεται από τη συνθήκη της Ρώμης ήδη και δεν έχει αλλάξει. Προστασία του περιβάλλοντος και του Γεωργού. Άρα δεν υπάρχει θέμα ως προς τους στόχους της ε, γεωργικής πολιτικής. Όντως, για τη γεωργική πολιτική δαπανούμε 54 δισεκατομμύρια το χρόνο. Μη λησμονούμε όμως ότι σε άλλες χώρες είναι πολύ πιο υψηλό το επίπεδο των δαπανών για τη γεωργική τους πολιτική. Ας κοιτάξουμε τις ε, αντίστοιχες τιμές για τις ΗΠΑ και με ΑΕΠ αντίστοιχο που έχει ξεπεράσει τα 80 δισεκατομμύρια σε ευρώ η δαπάνη για την ε, γεωργική τους πολιτική. Επομένως, ε, και αν κάνουμε και τις υπόλοιπες προσαρμογές με βάση το ΑΕΠ, το πληθυσμό κτλ, έχουμε τετραπλάσια ε, δαπάνη στις ε, Ηνωμένες Πολιτείες σχέση με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Γεωργία. Τώρα, στον αριθμό των γεωργών που δραστηριοποιούνται. Αυτό βεβαίως και παρουσιάζει πτωτική τάση. Έχει να κάνει με το εισόδημα που μπορούν να περιμένουν, με τη δραστηριότητα βεβαίως κατά κεφαλήν, ε, με την καινοτομία που πρέπει να ενισχύσουμε, για να βελτιωθεί η παραγωγικότητα, η οποία θα επιτρέψει στη συνέχεια και την καταβολή ψηλότερων αμοιβών στους γεωργούς. Η δουλειά μας είναι πολιτική, είτε εδώ είτε στο Συμβούλιο. Η δουλειά μας είναι να ορίσουμε στη μελλοντική μεταρρύθμιση της κοινής πολιτικής την επίτευξη ε, των στόχων κατά τρόπο που δεν θα στρεβλώνει τόσο, που δεν θα έχει δηλαδή τόσο ανετικέ συνέπειες ως προς το περιβάλλον, παραδείγματι. Αλλά αυτοί οι στόχοι δεν έχουν αλλάξει, όπως είπα, από τη συνθήκη της Ρώνη Κατά τα άλλα, συμφωνώ με την κυρία Αγγιλέρα, με το θεωρούμενο πλεονέκτημα του προτινόμενου εθνικού στρατηγικού σχεδίου γιατί βλέπω ότι κάποιες χώρες έχουν δυσκολίες προς και την διάρθρωση σε περιφερειακό επίπεδο αυτών των ε, σχεδίων. Και θα χρειαστούν ενδεχομένω ε, και δεκάδες, αν όχι περισσότερα, περιφερειακά προγράμματα. Ο κύριος Ανδρίο έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ζητώντα συγγνώμη για την ε, ολιγόλεπτη απουσία μου κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για άλλη μια, δουλειά, ε, για άλλη μια φορά για τη δουλειά που κάνετε από το Ελεκτικό Συνέδριο. Υπάρχουν κάποια σημεία και είναι σημαντικό πιστεύω να επιστρέψει η, ο σκοπός, η έννοια του σκοπού της εξυπηρέτηση ενός σκοπού στη γεωργία και η αξιοπιστία της. Και πρέπει να κοιτάξουμε και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου βεβαίως λέμε πως η κοινή πολιτική πρέπει να διατηρήσει το κοινό χαρακτηριστικό, πρέπει να αποφύγουμε την επαναθνικοποίηση. Και θα ήθελα να ρωτήσω πώς μπορεί να διευκρινιστεί αυτό, να εξατομικευθεί όταν μιλάτε για τα εθνικά σχέδια. Γιατί εγώ πιστεύω ότι όταν υπάρχουν πολλαπλοί στόχοι και πολλαπλά επίπεδα στόχων, ε, de facto αναπτύσσονται διαφορετικές πολιτικές δημόσιες πολιτικές. Εάν θέλουμε λοιπόν να έχουμε κοινή στόχευση στην κοινή τουρκική πολιτική, δεν μπορούμε να αφήσουμε τον προσδορισμό των στόχων στο εθνικό επίπεδο, χωρίς να ξαναγυρίσει στην εθνικοποίηση ή στην εθνική οργάνωση η γεωργική πολιτική. Έχετε εσείς εχετε εσει ιδέα συγκεκριμένη, πρακτική. Σε αυτό θα ήθελα κάποιε πιο συγκεκριμένες πληροφορίε. Και επίσης, Αναφέρεστε συχνά στην έκθεση, ενδιαφέρον μου φαίνεται, στη συγχρηματοδότηση. Απορρέει από την ε, πρόταση της Επιτροπής βεβαίω και μάλιστα αναφέρεστε στη συγχρηματοδότηση στα θέματα της οικολογικοποίησης, αφού η Επιτροπή με τις προτάσεις της αναφέρεται στα νέα eco eco-skins που θεωρείται σημαντικά και ε, υλοποιήσιμα με βάση μια ενισχυμένη ε, αιρεσιμότητα προς το περιβάλλον και την αποκατάσταση ενός γεωργικού ε, μοντέλου, το οποίο βεβαίως θα είναι προς το συμφέρον και θα ενδιαφέρει και τον ε, γεωργό να το υλοποιήσει. Αυτό το scheme, λοιπόν, βεβαίως πρέπει να το μελετήσουμε περισσότερο. Στη συγχρηματοδότηση ωστόσο, ε, και εδώ έγκυται η ευρωπαϊκή προσθεμένη αξία, θα πρέπει αυτή να καλύπτεται κατά 100% από το προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χρηματοδότηση λοιπόν του EcoScheme με τις αυστηρές προδιαγραφές που ορίζουμε και αναφέρθηκε επίσης ότι θα εξαρτηθεί και από το γεωργικό μοντέλο εάν αφήσουμε αυτή τη στιγμή τη γεωργία να κάνει επιλογές και δρόμους και με εξαφνιάζει ο Αλμπερτές ο οποίος έχει επανειλημμένος και με επιμέλεια επισκεφθεί τους Βραζιλιάνους παραγωγούς δεν νομίζω ότι είμαστε σε θέση, αγαπητέ Άλπερ, να τους ε, ανταγωνιστούμε. Μιλούμε για ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα εδώ και 50 χρόνια. Μα η παραγωγικότητα έχει οδηγήσει στο ότι το αριθμό των γεωργών. Και κυρίως σε ορεινές περιοχές, αλλά και σε πιο έφορες ε, περιοχές. Λοιπόν, ε, θα πρέπει να δώσουμε άλλου συσχετισμού ως προϋποθέσεις, ποιότητα τροφίμων, υγιεινή τροφίμων. Αν κοιτάξουμε τι συμβαίνει στις ΗΠΑ και το Μεξικό παραδείγματι με την παχυσαρκία που σχετίζεται με την ποιότητα των τροφίμων που καταναλώνονται. Με την με... με... Αντίπαλό μας την παγκοσμιοποίηση, εμεί πρέπει να εστιαστούμε στην υγεία, στο περιβάλλον και εκεί μπορούμε να μιλήσουμε για δημόσιες ενισχύσεις. Μπορούν οι δημόσιες ενισχύσεις να καλύψουν κάθε σημείο της γεωργικής παραγωγής. Δεν πρέπει να διερωτηθούμε σε αυτό, εάν υπάρχει δυνατότητα και πώς. Υπάρχουν τα ερωτηματικά, τα βλέπω και στην έκθεσή σας. Αλλά πρέπει να δώσουμε και απαντήσεις με ένα μοντέλο που θα επιλεγεί. Ένα μοντέλο που θα υπηρετεί και την επιστημιστική ασφάλεια, αλλά και την επιστημιστική κυριαρχία, το έχουμε πει πολλές φορές. Και αυτό μέσα σε μια ε, ανοιχτή θεώρηση με το βλέμμα στραμμένο σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ. Κύριος ε, Ευχαριστώ πολύ. Ακούμε τη μείωση του 22% των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Και δεν χρειάζεται κανείς να είναι σοφός για να καταλάβει ότι αν συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων θα είναι εξαιρετικά μικρός και θα είναι τεράστιες. Επομένως, κατά την άποψή μου όμως αυτό δεν θα έπρεπε να σε εκπλήσει. Βεβαίως ότι υπάρχει μείωση του αριθμού μάλλον λέγεται ότι υπάρχει μια ε, μείωση του αριθμού και ότι οι αγροτικέ εκμεταλλεύσει οι παραμένουν είναι μεγαλύτερε. Αυτό όμω εγγυάται μεγαλύτερο εισόδημα σήμερα ή στο μέλλον. Ή μήπω τελικά θα υπάρχουν ε, ελάχιστοι αγρότε οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα στην πραγματικότητα να ζουν από το εισόδημά του σε αντίθεση με την κατάσταση που είχαμε στο παρελθόν οι αγρότε να αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο τη τοπική οικονομία. Και προ τα εκεί θέλουμε να πάμε. Θα ήθελα να σας επισημάνω μια μελέτη παρόμοια η οποία είχε γίνει πριν από τις προηγούμενες διαπραγματεύσεις για την ΚΑΠ ε, τότε. Για το μέλλον της ΚΑΠ συζητούσαμε. Θα ήθελα να μου πείτε πώς την αξιολογείτε και αν θεωρείτε ότι ήταν... Ε, ε, ποια είναι η άποψή σας για αυτή. Κύριε Νίκολς, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω ότι έχω μια διαφορετική προσέγγιση στη συζήτηση. Πιστεύω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να ρωτήσουμε είναι τι περιμένουμε από τον Γεωργό. Τι περιμένουμε από την Γεωργία και από την αγροτική οικονομία και την οικονομία τροφίμων. Μετά από το σκάνδαλο που είχαμε με το κρέας των αλόγων, νομίζω ότι όλοι καταλάβαμε ότι το καλό φαγητό κοστίζει. Εάν κανείς δεν είναι δηλαδή διατεθειμένος να πληρώσει την ορθή, ε, το αντίτιμο, θα έχει τέτοιου είδους σκάνδαλα. Μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για το γεγονό ότι οι αγρότε και οι κτηνοτρόφοι σε ολόκληρη την Ευρώπη παράγουν ένα ικανοποιητική καλή ποιότητα προϊόν, το οποίο είναι σε σωστή τιμή. Δεν γνωρίζω κανέναν αγρότη ή κτηνοτρόφο ο οποίο να είναι εκατομμυριούχο, ή εν πάση περιπτώσει, αν γνωρίζω ορισμένου, δεν έβγαλαν τα λεφτά του από, από την αγροτική παραγωγή. Επομένως, τουλάχιστον στην περιοχή μου. Δεν είναι δυνατόν να φανταστώ μια μικρή ή μεσαία αγροτική εκμετάλλευση να επιβιώνει χωρίς την επιδότηση. Η τιμή που φτάνει στον τελικό καταναλωτή συμπεριλαμβάνει το κόστος για το, τους μεσάζοντες, το σούπερ μάρκετ κτλ. Το ερώτημα λοιπόν είναι ε, πώς θα μπορούσαμε να έχουμε μια μεσότερη σχέση με τον παραγωγό έτσι ώστε να τον ενισχύουμε καλύτερα. Άκου πριν ε, την αναφορά του συναδέλφου μήπω κρύβουν κάτω από τα, στρώματά του λεφτά οι αγρότες. Πιστεύω ότι αυτό ήταν ένας μύθος παλιός. Ίσως βέβαια συνέβη σε κάποιες χώρες τι οποίες δεν μπορούσε κανείς να εμπιστευτεί τι τράπεζες. Όμω εγώ βρίσκομαι στην Επιτροπή Αγροτικό ε, Γεωργίας ε, και ακούω επί χρόνια τα ίδια στοιχεία. Ότι αυξάνεται ο μέσο όρο ηλικία των αγροτών. Ότι μειώνεται ο ρυθμό των εκμεταλλεύσεων. Ε, κάποια στιγμή δεν πρέπει κανεί να αναρωτηθεί πού πάμε. Γιατί αυτέ οι τάσει συνεχίζουν. Δεν ανακόπτονται. Βεβαίω έχουμε αύξηση των τεχνολογικών λύσεων που μπορεί να βοηθήσουν. Μπορούμε να βρούμε άλλου τρόπου για να βοηθήσουμε του αγρότε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και η παραγωγή του να γίνει πιο αποτελεσματική. Αλλά όλα αυτά επίση κοστίζουν. Τελικά όμω πρέπει να δούμε ποια είναι το, τα έξοδα, πόσο, πόσο, ποιο είναι το κόστος που χρειάζεται έτσι ώστε μια εκμετάλλευση σήμερα να παραμένει ζωντανή, να παραμένει ανταγωνιστική και αποτελεσματική, όχι μόνο να είναι ανταγωνιστική στο εσωτερικό της Ένωσης, αλλά να μπορεί να ανταγωνιστεί και στην διεθνή αγορά. Ε, εκτός αυτού γνωρίζουμε ότι οι γρότες αυτή τη στιγμή έχουν να αντιμετωπίσουν μεγάλη βεβαιότητα. Δεν γνωρίζουμε, για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο τι θα συμβεί στο μέλλον, δεν γνωρίζουμε πού πάμε με τον Brexit. Ε, αυτό που ακούν οι αγρότες μας είναι ότι φέτος εντάξει του χρόνου βλέπουμε. Εγώ δεν θα ήθελα επίση σε καμία περίπτωση εξαιτία τη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πληγούν δυσμενώ αγρότε σε οποιοδήποτε άλλο μέρο τη ε, Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε ότι χρειάζεται, χρειάζονται επενδύσει. Πολλοί από τους γαλακτοπαραγωγούς σήμερα α, μου λένε ε, ότι χρειάζονται περισσότεροι, ότι ακούνε μάλλον από τους γιους τους, από τους νέους, να λένε ότι δεν θέλουν να έχουμε διευθυντεθειμένοι να συνεχίσουμε στην ίδια δουλειά, αν δεν υπάρξει περισσότερη αξιοποίηση της τεχνολογίας, αν δεν χρησιμοποιήσει ρομποτικές λύσεις, γιατί εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να δουλεύουμε όσο σκληρά δούλευε στο παρελθόν. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Στη Βραζιλία. Ξέρετε ότι έχουν δύο υπουργού για τα γεωργικά. Ένας ασχολείται με τις μεγάλε εκμεταλλεύσεις και ένας με αυτό που ονομάζουν κοινωνικές εκμεταλλεύσεις. Μια άλλη προσέγγιση. Κάπω ε, ε, μια διαφορετική προσέγγιση πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε κι εμείς. Όμω δεν γίνεται να συνεχίσουμε να επιτρέπουμε στους αγρότες, να τους επιτίθενται όλες οι μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις, όλες οι μεγαλύτερες δυνάμεις και ταυτόχρονα να τους ζητούμε να αντιμετωπίσουν όλο και μεγαλύτερη γραφειοκρατία, όλο και μεγαλύτερη πλημμυρίδα προϊόντων αγροτικών που έρχονται από όλες τις υπόλοιπε περιοχές του κόσμου και σε περιοχές τις οποίες σε καμία περίπτωση δεν τηρούνται τα ίδια πρότυπα ποιότητας ή περιβαλλοντικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα να τους ζητούμε να συνεχίσουν να είναι αγρότες και για τις επόμενες γενιές. Ευχαριστώ. Σράερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό που είπε ο κύριος Νίκολσον ε, με ευνηδίασε την περασμένη εβδομάδα ο κύριος Χαϊτεμά σε μια συνέντευξη στο ραδιόφωνο και είπε ότι οι γεωργοί δεν χρειάζονται άμεσες ενισχύσεις. Και οι γεωργοί έχουμε ακούσει πολύ συχνά ότι χρησιμοποιούν ε, τις νέες τεχνολογίες, χρησιμοποιούν τα ρομπότ. Και 80% των ε, Ολλανδών θα είχαν εγκαταλείψει τη γεωργική, είχαν εγκαταλείψει την γεωργική δραστηριότητα χωρίς τις άμεσες ενισχύσεις. Ε, εσείς στο ελεκτικό συνέδριο. Εξαρτώμαστε από τα στοιχεία που μας δίνετε για το δημοσιονομικό έλεγχο. Ο κύριος Δεκάστρο μίλησε για καινοτομία και είπε ότι είναι πολύ σημαντική η καινοτομία. Τι κάνουμε όμως για την καινοτομία. Χρειάζονται περισσότερα κονδύλια για να χρηματοδοτήσουμε την καινοτομία. Και τι γίνεται με τις μεγάλες γεωρικές εκμεταλλεύσεις. Είναι καινοτόμε. Ε, υπάρχουν στοιχεία για τις μεγάλες αυτές γεωρικές εκμεταλλεύσεις. Γιατί έχουν ένα μάνατζερ, ένα γενικό διαχειριστή που οργανώνει το διαγωνισμό στην Δανία που στην Ευρώπη για να προμηθεύονται με τις χαμηλότερες δυνατές τιμές. Αλλά πόσα κονδύλια λαμβάνουν αυτοί και πόσα οι απλή γεωργοί στα χωριά. Αυτά τα στοιχεία θέλω. θα πρέπει να εγγύψουμε στις μεγάλες εκμεταλλεύσεις, γιατί έχουμε από τη μια τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις και από την άλλη τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Αυτές βρίσκονται στην καρδιά της υπαίθρου και αυτές συντηρούν την υπαίθρο. Θα πρέπει πρώτα να συμφωνήσουμε τι εστί μεγάλη και τη μικρή γεωργική εκμετάλλευση. Γιατί και εκεί υπάρχουν διαφορές. Αλλά αν αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα δεν ξέρω πώς θα βρούμε προ... Ε, διέξοδο. Ο κύριος Χανιώτης, ο διευθυντής παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ή μάλλον η κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα αφήσω κατά μέρο τα θέματα τώρα σχετικά με τους στόχους, τις ε, πολιτικές επιλογές και τα υπόλοιπα στο συνάδελφο Χανιώτη. Θα ήθελα να πω δύο λόγια σε σχέση με, την, ε, με το τμήμα που αφορά την διαβεβαίωση από την ε, έρευνα, από την μελέτη αυτή και βεβαίως το μοντέλο που μπορεί να υλοποιηθεί. Νομίζω ότι μπορούμε να λάβουμε σημεία σημείο αφετηρία στην προηγούμενη συζήτηση για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης. Εκεί πολλοί είπατε ότι δεν έγινε απλούστευση, αλλά το αντίθετο, πε, περιπλάξε τα πράγματα. Και νομίζω ότι το πρόβλημα ε, της ΚΑΠ που είναι περίπλοκο είναι ότι χρειάστηκε να έχουμε γενικούς κανόνες και ε, κανόνες επιλεξιμότητας σε επίπεδο δικαιούχου, ενώ το νέο μοντέλο των αποτελεσμάτων αφήνει διακριτική ευχαίρεια στα κράτη-μέλη. Αυτά θα πρέπει να καθορίσουν τους κανόνες και να βρουν κανόνες και διατάξεις που προσαρμόζονται στην ιδιαιτερότητά του, στη δική τους πραγματικότητα, για να μην έχουμε ένα μοντέλο που να ταιριάζει, να εφαρμόζεται σε όλους. Οπότε... Ε, οι μεγαλύτεροι απορροφούν τα περισσότερα κονδύλια και οι κανόνες είναι ακατάλληλοι γιατί δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά όλων. Οπότε λέμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να θεσπίζουν τους κανόνες για τους δικαιούχους, ε, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες τους. Ε, φυσικά θα πρέπει τα μέτρα αυτά, οι διατάξεις αυτές να συνάδουν με, τον, ε, με τους ευρωπαϊκούς στόχους. Αυτά θα σας τα πει ο κύριος Χανιώτης. Ο κύριος Κάρσον είναι ο μόνος που μίλησε για το νέο, το delivery model. Η ιδέα δεν είναι στο μέλλον να σταματήσουμε τις βασικές ενισχύσεις ε, σε ένα γεωργό αν δεν υλοποιεί τους στόχους. Δεν είναι αυτό η έννοια του delivery model. Το θέμα είναι ότι οι στόχοι θα προσδιορίζονται σε εθνικό επίπεδο. Οπότε θα έχουμε μια νέα σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρατών μελών ε, στο νέο delivery model. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θέτει τους γενικούς στόχους και τα αποτελέσματα και θα λέμε τη σχέση μεταξύ δαπανών και ε, κρών, αλλά όχι σε επίπεδο μεμονωμένου γεωργού. Αυτό είναι αδύνατο για το μέλλον, γιατί φυσικά υπάρχουν και πολλοί εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τους μεμονωμένους γεωργούς. Τα κράτη-μέλη λοιπόν θα είναι υπεύθυνα αρμόδια για την υλοποίηση των στόχων, όχι οι μεμονωμένοι γεωργοί. Και οι διατάξει θα θεσπίζονται σε εθνικό επίπεδο, θα είναι εθνικέ διατάξει. Πάντω ε, χαιρετίζουμε αυτό το ενημερωτικό έγγραφο του ελεγκτικού συνεδρίου. Είναι μια πολύ θετική συνεισφορά για το νέο μοντέλο, το μοντέλο που θα στηρίζεται στα αποτελέσματα, το νέο delivery model και περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις και σχόλια ως προς αυτό. Ο κύριος Χανιώτης. Συνεχίζω λοιπόν την, την, τις προτάσεις της ε, να κάνω κάποια σχόλια για το γενικό προσανατολισμό ε, του εγγράφου. Το νέο μοντέλο αυτό έχει ως σημείο φετηρία στους στόχους. Αυτό είναι το delivery model που λέμε. και αυ... Ε, ρώτησε πριν ο κύριος Φλάναγκας που είναι το κοινό στην κοινή πολιτική. Έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις αλλά το κοινό της κοινή κοινής πολιτική πολιτικής έγκυται στους στόχους μας. Οι στόχοι δεν είναι μεμονωμένοι, δεν είναι ειδικοί, δεν αφορούν τη συγκεκριμένη γεωργική εκμετάλλευση, το συγκεκριμένο εισόδημα. Είναι μια ασφαλιστική δικλίδα για το γεωργικό εισόδημα και επιτρέποντα διαφοροποίηση στα κράτη-μέλη. Το ίδιο έγινε και για τις τιμές ε, παρέμβασης. Ε, ένα ε, δίκτυο ασφαλείας, ώστε τα κράτη-μέλη σε περίπτωση που μειώνονται οι τιμές έχουν ένα σύστημα για να χαλαρώνουν την πίεση σε επίπεδο γεωρική εκμετάλλευση, κρατώντα το γενικό πλαίσιο. Και αν κινηθούμε προς την κατεύθυνση των επιδόσεων, ε, των αποτελεσμάτων σε δείκτες που θα καταμετρούν τι τις επιδόσεις θα πρέπει να διευκρινίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε, τι επιδιώκουμε. Και το γεγονός ότι έχουμε τόσες ερωτήσεις για την εισοδηματική στήριξη μας δίνει την ευκαιρία να εξηγήσουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Καταρχήν, αυτή η μετατόπιση προς τα αποτελέσματα προϋποθέτει ε, να έχουμε σωστά στοιχεία. Χωρίς στοιχεία δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε δείκτες και να καταμετρήσουμε ή να αξιολογήσουμε τις επιδόσεις. Και βέβαια πολλές φορές ε, υπάρχει διάσταση για τα στοιχεία και τις γνώσεις και αν συμφωνούμε σε κάτι είναι ότι η γεωργία δεν είναι ένας κλάδος με ανθυρό εισόδημα. Αλλιώ δεν θα εξηγούσαμε τι στατιστικέ ή το γεγονό ότι έχουμε όλο και μεγαλύτερη έξοδο εργατικού δυναμικού από τη γεωργία. Με επίπτωση την αύξηση της παραγωγικότητας ε, του εργατικού δυναμικού και αυτή η έξοδος οφείλεται στις πιέσεις που οφείλεται, που οφείσταται ο γεωργικός κλάδος. Πολύ α, ε, καλό πράγμα η συζήτηση, αλλά εμείς 15 χρόνια συζητάμε το κατά πόσο ε, η, το επίκεντρο της κοινή γεωργικής πολιτικής αν θα πρέπει να είναι το γεωργικό εισόδημα, το εισόδημα της γεωργικής δραστηριότητα ή το εισόδημα γενικώ του της γεωργικής εκμετάλλευσης. Και ίσως έχουμε μια καλύτερη εξήγηση ε, για το γιατί γίνεται η διαφοροποίηση. Γιατί αυτό που προβλέπει η συνθήκη, φαίνεται και στο παράρτημα, είναι ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι κυρίως να επικεντρωθούμε στην αύξηση των αποδοχών των γεωργών. Και γιατί το λέω. Γιατί στόχος της κοινή γεωργικής πολιτικής δεν είναι να αντιμετωπίσει ε, ζητήματα που εμπίπτουν στην εθνική αρμοδιότητα. Και τα γεωργικά νοικοκυριά ε, έχουν σχέση με τη φορολογία που είναι εθνική πολιτική. Το συνταξιδοτικό σύστημα επίση είναι εθνική πολιτική και καθορίζει το ποιοι θα παραμένουν και ποιοι θα φύγουν. Επίση, το κληρονομικό δίκαιο είναι εθνική πολιτική. Αγορές ακινήτων επίσης είναι εθνική πολιτική. Και το έχουμε πει επανειλημμένω και εδώ και στο δικαστήριο. Η κατηγορία ότι οι άμεσε ενισχύσει επηρεάζουν αρνητικά τι τιμέ των αγεών είναι ανεδαφική και ανεδαφικές και σας καλώ να εξετάσετε πρόσφατα δημοσιεύματα της Ευρωπαϊκή Επιθεώρηση Γεωργική οικονομία, που δικαιολογούν αυτά που σα λέμε εδώ και χρόνια. Και πρόκειται για πρόσφατο δημοσίευμα, σα το συστήνουμε. Δεν επηρεάζουν οι βασικές ενισχύσει αρνητικά το επίπεδο των Τη τιμής της γης. Και όταν μιλούμε για στόχευση, τι θέλουμε να στοχεύσουμε, σε τι, στη γη ή στον μεμονωμένο αγρότη. Γιατί αν θέλουμε να στοχεύσουμε στον μεμονωμένο αγρότη, χρειαζόμαστε ολόκληρο στρατό που να ελέγχει την παραμικρή λεπτομέρεια της γεωργικής δραστηριότητας. Αν όμως επικεντρωθούμε στη γεωργική επιφάνεια, στη γεωργική έκταση, στη γεωργική εκμετάλλευση, συνδυάζουμε καλύτερα τις ε, οικονομικές και τις περιβαλλοντικές δραστηριότητε του Γιώργου. Και επίσης ε, αναφέρουμε κάτι που συχνά θέλουμε να αποφύγουμε. Το γεγονό, δηλαδή ότι μπορεί να έχουμε τις ε, εκμεταλλεύσεις με τις καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις που δίνουν όμω ε, οικονομικά προσοδοφόρες για να παραμείνουν στην αγορά. Ενώ έχουμε άλλε γεωργικές εκμεταλλεύσεις με καλέ οικονομικές επιδόσεις αλλά με χαμηλέ περιβαλλοντικέ επιδόσεις. Και αυτό που είδαμε σε όλε τι συζητήσει που είχαμε κατά τι δημόσιε διαβουλεύσεις για το μέλλον τη κοινή γεωργική πολιτική είναι ότι όλα τα θετικά παραδείγματα που εντοπίσαμε και που δείχνουν πώς μπορούμε και να επιτρέψουμε περισσότερη επικουρικότητα και να απλουστεύσουμε τις πολιτικές, αυτό προέρχεται κυρίως από τον εξυγχρονισμό των βέλτιστων πρακτικών. Και ταυτόχρονα έχουμε αύξηση και των οικονομικών και των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Έχουμε ένα πάνελ βέλτιστων πρακτικών που καλέσαμε στη ε, πρόσφατη διάσκεψη του Δεκεμβρίου και από εκεί θα βρείτε πολλές πληροφορίες για το θέμα αυτό. Και αυτός είναι ένας τομέας που πιστεύουμε έχει τη δυνατότητα και να έχει σαφώς στοχοθετημένη προσέγγιση στο μέλλον. Και τέλος, όταν μιλούμε για τους στόχους, αυτό που θα δείτε στην μελέτη επιπτώσεων των προτάσεων και αυτό που είπαμε ήδη στην ανακοίνωση, είναι η προσπάθειά μας να υιοθετήσουμε ισορροπημένη, πολύ ισορροπημένη προσέγγιση με ανάλογα με τι τρει διαστάσει τη κοινή γεωρικής πολιτική. την οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική. Σε ό,τι αφορά την οικονομική και την περιβαλλοντική διάσταση τη κοινή γεωρικής πολιτική, έχουμε μια μελέτη επιπτώσεων και φαίνεται ότι το οικονομικό σκέλος έχει καλύτερε επιδόσεις από το περιβαλλοντικό. Τίποτα δεν είναι τέλειο, αλλά τίποτα δεν είναι και χάλια. Σίγουρα τα οικονομικά αποτελέσματα της ΚΑΠ είναι πιο θετικά από τα περιβαλλοντικά. Στην κοινωνική διάσταση είναι που έχουμε ένα κενό και που καλύπτεται την πρόσφατη μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας με βάση μια πλούσια βάση δεδομένων που εξετάζει το επίπεδο βασικής ενίσχυσης, πρώτο και δεύτερο και τις τυχικές περιφτώχειες σε επίπεδο ΝΑΤΣ 3. Όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι η ΚΑΠ είναι παρούσα παντού με θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη, την ε, απασχόληση και θετική μείωση ή θετική σύνδεση με τις αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις. Θετική επαφή με τις αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις. Γενικώ χαιρετίζουμε την επισκόπηση, αλλά εντοπίσαμε και κάποιους κανόν, κλάδους όπου θα πρέπει να προσδιορίσουμε τους στόχους μας. θα προτείνουμε καλύτερη καταμέτρηση αυτών των στόχων και θα αναφέρουμε και την προστιθέμενη αξία της κοινή γεωρικής πολιτικής. Έχουμε όλο και λιγότερο χρόνο. Ο κύριος Φίλικ αρχίζει και ανησυχεί. Μισό λεπτό Χόισλινγκ και οι υπόλοιποι. Μισό λεπτό καθένας. Μας λέτε πώς θα λειτουργήσουν αυτά τα ωραία καινούργια πράγματα. Περιμένω όμως με ενδιαφέρον να δω στην πραγματικότητα τι θα συμβεί, γιατί είναι πολύ εφηρημένες αυτές οι υποσχέσεις, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω συγκεκριμένα. Ε, λέτε ότι η ρύθμιση των ποσών θα γίνει μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει σχέση με τους γεωργούς. Και μετά στη δεύτερη φράση μας λέτε ότι... Ε, δεν είναι όλα τα πράγματα στραβά στην Ευρώπη. Μα κάνετε κάτι περισσότερο, εν πάση περιπτώσει, για να λυθούν τα προβλήματα και κάτι ακόμη Φαντάζομαι θα ξέρετε τον μύθο με τον Αϊτό και το, και το λαγό. Είναι άνισος ο αγώνας δηλαδή. Ο Επίτροπος σήμερα χαιρετίζει μια νέα συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με το Μεξικό. Δηλαδή βάζουμε στην ίδια ζυγαριά τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές με τις προδιαγραφές των άλλων κρατών του κόσμου. Βραζιλία, όπου έχει πάρει μια νέα ε, τελείως έννοια η οικογενειακή εκμετάλλευση. 180.000 εκτάρια η οικογενειακή εκμετάλλευση στη Βραζιλία. Με αυτούς θα ανταγωνιστούμε. Με συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών δεν μπορούμε να έχουμε κανένα αποτέλεσμα ισοφελός μας από αυτά. Πρέπει να τα βάλουμε όλα στη ζυγαριά για να φέρει αποτελέσματα αυτή η πολιτική. Κύριος Δέσης. Μισό λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σπάνια συμφωνώ με τον Μάρτιν Χόισλινγκ, όμως εδώ σχεδόν, σχεδόν συμφωνούμε. Δεν θα προκύψει λιγότερη γραφειοκρατία από τα όσα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απλώς θα μεταφερθεί στα κράτη-μέλη. 16 δε τα κρατήρια της Γερμανίας, καταλαβαίνετε. Ανταγωνισμός και στρέβλος ανταγωνισμού μεταξύ των ε, κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Γερμανία ενδεχομένως μεταξύ των κρατηδίων της Ομοσπονδιακής χώρας. Και νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς να πει ότι και 50% των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής περισσεύει, αλλά μένουν στις θέσεις τους για να, μάλλον για να μείνουν στις θέσεις τους προγραμματίστε, σχεδιάστε μια γεωργική πολιτική που θα δικαιολογήσει την παραμονή τους. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι λύση για τη γεωργική πολιτική. Από αυτά που ακούμε και από το Ελεγκτικό Συνέδριο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πιο πολύ φοβούμε την Επιτροπή παρά το Ελεγκτικό Συνέδριο. Έχω την αίσθηση ότι ό,τι έκανε η Επιτροπή ήταν αρνητικά. ό,τι και να κάνει αρνητικά το κρίνουμε. Όχι, κάπου θα πρέπει να α, συναντηθούμε. Δεν μπορεί να το α και το αντίθετο του α είναι εξίσου αρνητικά. Είναι σημαντικό να έχουμε συζήτηση και επιστημονικό χαρακτήρα, αλλά να μην περιοριστούμε στη θεωρητικολογία. Κύριε Φιγκερέντο, δεν χρειάζεται να απαντήσετε διεξοδικά σε όλες τις ερωτήσεις. Παρακαλώ σύντομα και συνοπτικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής για τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ επίσης και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις παρατηρήσεις τους. Θα ξεκινήσω από μία απάντηση δική μου και με την άδειά σας κύριε Πρόεδρε θα δώσω το λόγο και στον συνάδελφο για να προσθέσει ορισμένα στοιχεία. Πρώτα απ' όλα. Όλα όσα θα πω τα λέω με, τον, με πλήρη σεβασμό στο ρόλο σας. Εκπροσωπείτε τους Ευρωπαίους πολίτες. Εσείς θα καθορίσετε τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και οτιδήποτε πω το λέω με πλήρη σεβασμό στον σημαντικό και απολύτως ε, κρίσιμο ρόλο σας. Ακόμα και αν ασκήσω κριτική. Πρώτα απ' όλα, κάποιο ανέφερε ότι αυτό, ότι αυτό το έγγραφο είναι πολιτικό. Δεν είναι ένα πολιτικό έγγραφο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο επαναλαμβάνουμε παρατηρήσεις, ευρήματα, ε, συμπεράσματα στα οποία είχαμε καταλήξει σε προηγούμενες εκθέσεις τις οποίες είχαμε αποστείλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι συστάσεις, παρατηρήσεις, οι οποίες βασίζονται στα ευρήματά μας από, από όλα τα κράτη-μέλη, όπου γίνονται επιτόπιες επισκέψεις των ελεκτών του ε, ελεκτικού συνεδρίου. Η κοινή αγροτική πολιτική είναι μεγάλη δαπάνη, ή μικρή. Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ. Δεν είναι ο ρόλος του ελεγκτικού συνεδρίου να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Το μόνο πράγμα που μπορεί να πει το ελεγκτικό συνεδρίο είναι να κρίνει ή μάλλον να επισημάνει ότι η ΚΑΠ αποτελεί το 39% των εξόδων του Γενικού Προπολογισμού της Ένωσης. Το ένα αυτό είναι πολύ λίγο, με όλο το σεβασμό, είναι δικιά σα απόφαση, είναι δικιά σα ε, θέση, γνώμη. Εμεί δεν μπορούμε να έχουμε μια συγκεκριμένη θέση από αυτό. Κάποιοι είπαν δεν χρειαζόμαστε περισσότερα στατιστικά στοιχεία. Υπό μία έννοια ίσως να συμφωνώ. Γιατί μπορεί να θεωρώ ότι χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία, για παράδειγμα όσον αφορά το αγροτικό εισόδημα γιατί εδώ εντοπίζω κάποιες, κάποια προβλήματα, κάποιες αδυναμίες. Συνολικά όμως, συμφωνώ, δεν χρειάζεται να αποκτήσουμε ακόμα περισσότερα στατιστικά στοιχεία. Όμως αυτό που ζητούμε από τον συνομοθέτη είναι να προσέξει τα στοιχεία, τα στατιστικά, τα αριθμητικά στοιχεία όταν θα εγκρίνει τη νέα ΚΑΠ. Με λίγα λόγια, μην βασιστείτε σε ε, προκαταλήψεις, σε μια εικόνα που την οποία έχετε ήδη ε, ε, ε, διαμορφώσει, αλλά κοιτάξτε τα πραγματικά δεδομένα. Πού τα, από πού τα συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα. Για όλα τα στατιστικά στοιχεία απο που τα συλλεγουμε αυτα τα δεδομενα για ολα τα στατιστικα στοιχεια που αναφερουμε στο έγγραφο αυτό, έχουμε αναφέρει και την πηγή. Εάν δεν ε, του, βρίσκεται την παραπομπή αρκετά ξεκάθαρη, μπορούμε να τη διευκρινίσουμε περαιτέρω. Γνωρίζουμε όμω όλε τι πηγέ των στοιχείων μα και θα αναφερθεί περισσότερο σε αυτό το θέμα και ο συνάδελφο. Για το ζήτημα τη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, που είναι και αυτό ένα ζήτημα που εσεί αναδείξατε. Το ελεκτικό συνέδριο δεν έχει έναν δικό του ορισμό Τη προστιθέμενης αξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν αποτελεί αρμοδιότητα του ελεγκτικού συνεδρίου να ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο ασκούνται οι πολιτικές στην Ένωση. Ακόμα και σε προηγούμενες εκθέσεις μας σε σχέση με τη μελλοντική κατανομή των πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είπαμε ότι χρειάζεται να εγκριθεί από τους συνομοθέτες ένας ορισμός πιο ξεκάθαρο για το τι συνιστά ευρωπαϊκή προστεθέμενη αξία. Δεν είναι δουλειά του, Ευρωπαϊκού, του Ελεκτικού Συνεδρίου να καταλήξει σε αυτόν τον ορισμό. Επισημαίνουμε όμως ότι εσείς, οι συνομοθέτες, πρέπει να καταλήξετε σε έναν ξεκάθαρο ορισμό. Άκουσα επίσης με την κριτική ότι ίσως να είμαι υπερβολικά αισιόδοξο για αυτό το νέο delivery model ή υπερβολικά αισιόδοξο για αυτά τα εθνικά στρατηγικά σχέδια. Εγώ δεν είμαι ούτε αισιόδοξο ούτε απεσιόδοξο. Περιμένω να δω συγκεκριμένε προτάσει για να δω τελικά πώς θα καταπίζονται αυτά τα εθνικά στρατηγικά σχέδια, Ποιο θα είναι ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή τη διαδικασία, ποιο θα είναι όλο το πλαίσιο με βάση το οποίο θα αξιολογούμε την εφαρμογή της ε, κοινή αγροτικής πολιτικής και τις επιδόσεις μας τα επόμενα χρόνια. Η προσέγγιση που έχω είναι περιμένουμε να δούμε τι θα έρθει. Δεν είναι αισιόδοξο αυτό, δεν είναι ούτε απεσιόδοξο. Το ερώτημα το ποιο, ποια θα πρέπει να είναι, εάν ο στόχος της ΚΑΠ θα πρέπει να είναι μάλλον η, δημο, η χρήση δημοσίων δαπανών, η, υπέρ των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, υπέρ της γεωργίας. Αυτό και πάλι δεν είναι ένα ερώτημα που εμείς μπορούμε να απαντήσουμε. Στο έγγραφο μας επισημαίνουμε ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικοί μηχανισμοί που μπορούν να αξιοποιηθούν για την εντόπιση των προβλημάτων των αγροτών και αυτών των περιοχών και η ΚΑΠ είναι ένας από αυτούς τους μηχανισμούς όμως στην έκθεση για το βασικό καθεστώς ενίσχυσης. διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια, υπάρχει μια φθήνουσα τάση ε, του βασικού καθεστώτος ενίσχυσης. Και αναφέρθηκα επίση εντάχει στο περιβάλλον στην παρουσίασή μου, αλλά στο έγγραφο θα βρείτε ένα ολόκληρο κεφάλαιο για το θέμα, στο οποίο εξετάζουμε τη συνεισφορά της κοινή αγροτικής πολιτικής στην προστασία του περιβάλλοντος. Και με την άδειά σας κύριε Πρόεδρε, τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον συνάδελφό μου για πέντε λεπτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Για το θέμα του περιβάλλοντος. Είναι σχετικά σύντομο το έγγραφο, 30 σελίδες, επομένως δεν έχει δώσει πολύ χώρο στο περιβάλλον. Αναφερόμαστε όμως στις κύριες προκλήσεις για το περιβάλλον στην Ευρώπη. Και λέμε ότι δεν αρκεί η πρόοδος στις περιβαλλοντικές κυκλούς, στους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους της ΚΑΠ. Και λέμε επίσης ότι η ΚΑΠ θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί ακόμη περισσότερο με άλλους σημαντικούς στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων βεβαίως το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή. Άρα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης ακόμη. Και θα ήθελα σύντομα να πω για τα δεδομένα και τις στατιστικές. Συμφωνούμε νομίζω ότι είναι πολλά τα δεδομένα που κυκλοφορούν. Το πρόβλημα όμως αντιμετωπίζουμε είναι η ποιότητα των δεδομένων, η αξιοπιστία τους, η χρησιμότητά τους για τους στόχους της ΚΑΠ. έτσι ώστε και να μεταφράζονται σε πιο λειτουργικούς όρους στην νομοθεσία. Γιατί βλέπουμε ότι τα αποτέλεσματα δεν είναι αυτά που θα θέλαμε, δεν είναι λειτουργικά. Χρειαζόμαστε ένα πιο συνεπές, ένα πιο λογικό σύστημα, καλύτερη ποιότητα και ίσως και πρόσθετα στοιχεία σε κάποιους τομείς της πολιτικής. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούμε για τις τάσεις, της ισοδημοτικές, είναι τα δεδομένα που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις ε, μελέτες της Eurostat, TN, και έχουμε σημειώσει και σε άλλες εκθέσεις ότι υπάρχουν ε, κάποια προβλήματα σε σχέση με την ποιότητα των δεδομένων, αλλά είναι τα καλύτερα που έχουμε στη θέση μας και γι' αυτό και τα χρησιμοποιούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Σέρμαν. Ο Πρόεδρος, χωρίς μικρόφωνο. Ναι, ήταν μεγάλη χαρά και για μας Είναι μεγάλο το έργο που έχετε και πολλές ευθύνες. Είμαστε βεβαίως σε μια εξελίξη συζήτηση, δεν έχει τελειώσει εδώ η συζήτηση, θα διατηρήσουμε την επαφή. Σας ευχαριστώ προς το παρόν. Κλείνουμε εδώ αυτό το σημείο και πρέπει να πω ότι το να δουλεύουμε χωρίς περιορισμούς χρόνου μερικές φορές ε, πράγματι μας ε, δίνει πολύ καλή ποιότητα δουλειά. Σε ευχαριστώ λοιπόν και εσάς και όλους όσοι έλαβαν το λόγο και τους εκπροσώπους αυτής της Επιτροπής. Και περνούμε στον προπολογισμό 2019, σημείο 9, εντολή για τριμερή διάλογο με τον κύριο Ραμόν Λουίς Σίσο. Ε... Πανέμορφο ονοματεπώνυμο. Αρμόδια κατ' ουσία επιτροπή είναι Επιτροπή Προπολογισμών. κυρία Δανιέλ, ο κ. Δανιέλ Βιώτη είναι αρμόδιος κατ' ουσίαν, εισηγητής. Επίσης, θα περιλαμβάνει η έκθεση της ε, Επιτροπής Προπολογισμών την ψήφισμα με την πρώτη αντίδραση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο σχέδιο προπολογισμού του 2009 που θα υποβάλει στα τέλη Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι επιμέρους επιτροπές έχουν δυνατότητα να καταθέσουν γνωμοδότηση μέχρι τις 21 Ιουνίου στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και σε τα πλαίσια αυτής της διαδικασίας ε, και εκ μέρους Επιτροπής Γεωργίας τη γνωμοδότηση θα εκπονήσει ο κύριος ε, Ραμόν Λουίς Βαλκάρσελ Σίσο. Κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για το λόγο που μου δίνετε και ευχαριστώ και για τα ευγενικά σας, ε, ευγενικά σας σχόλια ως προς το ονοματεπώνυμό μου ή τα επώνυμά μου που προέρχονται και από τη πλευρά του πατρός και της μητρός. Νομίζω ότι είναι σημαντική αυτή η γνωμοδότηση για την Επιτροπή Γεωργίας γιατί αναδεικνύει τα κέρια θέματα και το ρόλο της, ε, σημαντικό ρόλο της Γεωργίας για την επίτευξη των κοινοτικών στόχων. Επίση, υποστηρίζει την απαραίτητη σταθερότητα του γεωργικού προπολογισμού στην οδηγία και είναι κατά οποιασδήποτε περικοπής και αυτό το λέμε καθαρά και εξάστερα. Ε, είναι σημαντικό αυτό το θέμα τη διασφάλιση του γεωργικού προπολογισμού, λαμβάνοντα υπόψη τι τεράστιε αστάθειε τιμών που έχει υποστεί ο γεωργικό τομέα κατά τα τελευταία έτη. Επίση, το σχέδιο γνωμοδότηση. Ε, ε, ε, ε, επισημαίνω και πάλι την ανάγκη υιοθέτηση μέτρων για να ε, αντιμετωπίσουμε ή να αντισταθμίσουμε τα αρνητικά αποτελέσματα του ρωσικού εμπάργου. Και θέλουμε να επεκταθούν οι, τα μέτρα υποστήριξης ε, που κανονικά λήγουν στις 30 Ιουνίου του 2018, γιατί το εμπάργο εξακολουθεί να επηρεάζει αρνητικά τις ευρωπαϊκές εξαγωγές. Επίσης, ε, τονίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει την πιθανότητα αυτά τα ε, έκτακτα μέτρα να μετατρέψει σε διαρθρωτικά μέτρα, γιατί δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ρωσία έχει καμιά πρόθεση να άρει το εμπάργο της. Το αντίθετο. Επανέρχομαι τώρα στο κείμενο της γνωμοδότησης. Ε, κατά κάποιο τρόπο έκανα σκόπιμο να προκαταλάβω κάπως τις συζητήσεις που θα έχουμε στα πλαίσια της μελλοντική μεταρρύθμισης της κοινή γεωρικής πολιτικής. Για παράδειγμα, εκφράζω ε, την σημασία που έχει η εξέταση ενός αποθεματικού κρίσης με πολιτική χαρακτήρα, άσχετα από, αποσυνδεδεμένο από τις βασικές ενισχύσεις, ε, ε, επιδεικνύοντας σε απαραίτητη πολιτική βούληση για, τις, ε, για το αποθεματικό αυτό που θα πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένο από τις άμεσες πληρωμές. Επίσης, καλό τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τα μέτρα στήριξης για τους νέους για να εξασφαλιστεί η ηλικιακή ανανέωση στη Γεωργία και εκφράζω την τον προβληματισμό μου και την ανησυχία μου για τις πιθανότητες που μπορεί να έχει για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στον προϋπολογισμό το 2019 μια ενδεχόμενη αποτυχία των διαπραγματεύσεων του Brexit. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της γνωμοδότησής μου που επικεντρώνονται στα σημαντικότερα κατά τη γνώμη σημεία για την Επιτροπή Γεωργίας και είμαι πρόθυμος να εξετάσω τις τροπολογίες σας. Πιστεύω ότι χάρη στην εργασία μας θα καταλήξουμε στο καλύτερο δυνατό κείμενο και περιμένω τα σχόλιά σας για να το εμπλουτίσουμε όσο γίνεται. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και σας κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κύριε Παλκάρσελ. Πρώτος ζήτησε το λόγο ο κύριος Μάρκ Ταραμπέλα. Πρόεδρε, ευχαριστώ δεν εκπροσωπώ τον εαυτό μου. Ο κύριο Δερανό μου ζήτησε να λάβω το λόγο εκ μέρου του, καθώ είναι ο σκιώδη των Σοσιαλιστών Δημοκρατών. Στην πρώτη παράγραφο θα ήθελα να προσθεθεί η αναφορά στην κοινωνική ισορροπία. Στην παράγραφο 2 δείχνουμε μόνο τη σταθερότητα του προπολογισμού τη Γεωργία, αλλά και τη διατήρηση στην τρέχουσα τιμή του προπολογισμού, αλλά και η θέλη μου αναφορά στις ε, εμπορικές συμφωνίες οι οποίες ε, οδηγούν πάντα σε αβαρία την γεωργία με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαπραγματεύση αυτή τη στιγμή. Στην πέμπτη παράγραφο δεν θέλω να γίνει αναφορά στο Brexit, ότι δεν πρέπει να επηρεάσει τον προπολογισμό του 2019 αφού το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευθεί να τιμήσει τις προσχέσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του τελευταίου πολίτου του δημοσιονομικού πλαισίου. Στην έκτη παράγραφο μπορούμε να συμφωνήσουμε σε σχέση με, το, με τα ελλείμματα και τα κενά, τα χάσματα που παρουσιάζει το ταμείο κρίσεω που έχουμε αυτή τη στιγμή, γιατί πρέπει να δώσει λύσει σε γεωργικέ κρίσει και πρέπει να έχουμε και ένα πρόγραμμα αντικυκλικό και στην 7η παράγραφο, την οποία βρίσκει εξαίρετο ο κύριος Δενανό. Θα ήθελα να προσθέσει και τις καλλιέργειες οι οποίες έχουν θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, όπως σε παραδείγματι της καλλιέργειας οσπρίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως ζωοτροφή, Αυτά ήθελε ο κύριος Δενανού να συμπληρωθούν στο κείμενο. Ζητώ συγγνώμη, μια και μια μικρή καθυστέρηση. Θα πρέπει να αποχωρήσω μέσω σε μια άλλη συνεδρία, στην οποία πάλι θα φτάσουμε καθυστέρηση. Με περιμένουν όμως και βεβαίως θα σημειώσουμε τα όσα έχει να πει στις απαντήσεις του εισηγητή. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Ταραμπέλα. Κυρία Κατάιναν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εκ μέρους της Άλτε θα ήθελα να ευχαριστώ τον εισηγητή για την ισορροπημένη ε, του έκθεση. Έχει λάβει υπόψη πολλά ζητήματα, σημαντικά ζητήματα, την υποστήριξη των νεαρών γεωργών, του μέλλοντος δηλαδή της γεωργίας και συμφωνώ με τον εισηγητή ότι ο γεωργικός προϋπολογισμός δεν αντέχει περικοπές υπό τις τρέχουσες συνθήκες. Οι γεωργοί έχουν δει του γεωργικού του εισοδηματός του είναι το 40% σε σχέση με τους λοιπούς τομείς. Η το εμπάρκο σε σχέση με τη Ρωσία, απαγορεύσεις εισαγωγών ε, πρέπει να ε, συνεχιστεί και τι αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα στην Φινλανδία ε, και τις χώρες της Βαλτικής που δεν έχουν μπορέσει να βρουν εναλλακτικέ αναφορέ, αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα προβλήματα που ταλανίζουν τους ε, γεωργούς. 370.000 τόνους είχαμε πριν από μερικά χρόνια σε σκόνη γάλακτος, ε, που όμως τελικά ρευστοποιήθηκε και έτσι αναγκάζονται πλέον οι γαλακτοπαραγωγοί να αποχωρήσουν ε, από τον τομέα ή να δεχθούν πολύ χαμηλές τιμές γάλακτος. 5,2 σεντ μείωση είδαν η παραγωγή μπορεί αυτό να οδηγήσει και στο τέλος του τομέα του γάλακτος στη Φινλανδία. Πρέπει λοιπόν να αναστήσουμε νέες λύσεις χωρίς προκαταλήψεις, με πνεύμα ανοιχτό. Τώρα που έχει καταργηθεί η στο γάλα, πρέπει ο κάθε παραγωγός να βρει τις δικές του λύσεις για την παραγωγή και σε λίγους τομείς μπορεί κανείς να, περι... να τηρήσει τα εθελοντικά ε, συστήματα αυτοπεριορισμού. Πρέπει να βρεθούν νέες λύσεις, πρέπει να έχουμε υπόψη της, τη ζημιά που μπορεί να φέρει το νέο σύστημα στην ε, γαλακτοπαραγωγή και μόνο με μεταρρύθμιση της κοινής πολιτική πολιτικής μπορεί να έχουμε καλύτερη διαχείριση κινδύνου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Σιβιέγας. Ευχαριστώ. Δεν πρόκειται να επαναλάβω τα σχόλια των προελισσάντων γιατί συμφωνώ με πολλά από αυτά. Θα ήθελα να υποστηρίξω πόσο σημαντικό είναι το θέμα της, του γεωρικού εισόδηματος. Αυτό θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της κοινή γεωρικής πολιτικής. Αυτό θα είναι το σημαντικό σημείο και ο βασικός μας προσανατολισμός. Γι' αυτή, αυτό το γεωρικό εισόδημα, πέραν το ότι ΚΑΠ αντιπροσωπεύει μεγάλο μερίδιο του κοινοτικού προϋπολογισμού και παρά τους λόγους και τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται για να κατηγορήσουμε το υπερβολικό κατά τη γνώμη μερίδιο της ΚΑΠ στον προπολογισμό, ε, οφείλουμε να διαπιστώσουμε ότι το γερικό εισόδημα εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλότερο από το εισόδημα εργαζομένων σε άλλους τομείς ε, της οικονομίας. Κάτι που ε, είναι πραγματικά αξιοθρύνητο και δεν μπορούμε να το καταλάβουμε κιόλα. Οπότε θα πρέπει να μιλήσουμε για το εισόδημα από ποσοτική σκοπιά. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αυξήσουμε το γεωργικό εισόδημα. Γιατί χωρί εισόδημα δεν θα προσελκύσουμε νέου αγρότε στην γεωργία. Και δεν πρόκειται ε, που δεν είναι να αντιστρέψουμε αυτή την κατεύθυνση τη εγκατάλειψη. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε δίκαιε τιμέ παραγωγή, ώστε να είναι προσοδοφόρα η γεωργική δραστηριότητα. Και από αυτήν την άποψη είναι, είναι εμφανέ ότι στην παρούσα κατάσταση ε, τα μέτρα και οι μηχανισμοί που έχουμε δεν έχουν αποφέρει καρπούς και προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε το, το σύστημα των ποσοστώσεων που για πολλά χρόνια επέτρεψε διατήρηση των τιμών σε συγκεκριμένα επίπεδα. Τώρα έχουν ε, σε, σε, επιδείξει κατακόρυφη πτώση, κάτι που φάνηκε στις τιμές του αποβουτυρωμένου γάλακτος στο σκόνη. Και όχι μόνο δεν έχουμε αύξηση του γεωρικού εισοδήματο, αλλά αντίθετα, μείωση. Επίση, να ληφθεί υπόψη μεγάλη αστάθεια, μεγάλη διακύμαση των τιμών γεωργικών προϊόντων. Και καλό θα ήταν να κατευθύνουμε τη συζήτηση για να κάνουμε μια διαφοροποίηση των παραγόντων τη αστάθειας των τιμών. Έχουμε τους, ε, τον περιβαλλοντικό, τον υγειονομικό κίνδυνο, αλλά αυτή η, η αστάθεια, η αβεβαιότητα των τιμών δεν οφείλεται σε, ούτε σε υγειονομικό κίνδυνο, ούτε σε κλιματικό ή περιβαλλοντικό κίνδυνο. Πρόκειται για πολιτικό κίνδυνο. Το εμπάργο της Ρωσίας, για παράδειγμα. Η δασμολογική της ρωσιας για παραδειγμα η δασμολογικη πόλεμοι που προδιαγράφονται. Οι εμπορικές συμφωνίες. Αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν την εξαιρετική διακύμαση των τιμών, την τεράστια στάθεια των γεωργικών τιμών. Και από τη στιγμή που υπάρχει αυτό ο πολιτικός κίνδυνος, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η τεράστια στάθεια των τιμών που οφείλεται και απορρέει από πολιτικές που εφαρμόζουν τα κοινοτικά θεσμικά όργανα, τότε θα πρέπει ο κοινοτικό προπολογισμό. ο προπολογισμό τη ΚΑΠ να αναλάβει το κόστος και τις συνέπειες των πολιτικών μέτρων που ελήφθησαν και που επηρεάζουν την καταβαράθρωση του γεωρικού εισοδήματο και την καταβαράθρωση των γεωρικών τιμών. Θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε τα απαραίτητα ταμεία και τα, να βρούμε τα απαραίτητα κονδύλια ώστε να αντισταθμίσουμε αυτή την απώλεια των εισοδημάτων και να αποφύγουμε μια εκατόμβη τη γεωργία. Επίση θα πρέπει να γίνει μια διαφοροποίηση των κινδύνων που επηρεάζουν αυτή την αστάθεια των τιμών και να διαχωρίσουμε τον πολιτικό κίνδυνο από του υπόλοιπου που μπορεί να είναι κλιματική, περιβαλλοντική ή υγειονομική. Αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο κοινοτικός προϋπολογισμός θα πρέπει να αντισταθμίσει την απώλεια εισοδήματο στους γεωργούς σε περίπτωση που ε, λόγω εμπορικής συμφωνίας με το Μερκοσούρ και καταβαράθρωση στον τιμό του κρέατος θα πρέπει ο κοινοτικός προϋπολογισμός να αντισταθμίσει αυτή την απώλεια. Δεν φταίνει οι κτηνοτρόφοι ούτε έχουν τη δυνατότητα μόνοι τους να αντιδράσουν και να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους πολιτικούς κινδύνους. Ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον Διευθυντή τον κύριο Χάισλερ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα δώσω μια γενική φύσεω απάντηση αυτή, γιατί γνωρίζετε ότι το πολιετέ δημοσιονομικό, μάλλον το προϋποδοσή μα για τον προπολογισμό θα έρθει ε, τέλη Μαΐου και τότε τα πράγματα θα είναι πιο ξεκάθαρα. Στον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις, το επίπεδο θα παραμείνει σταθερό κατά τη διάρκεια του 2019 με, μικρή, με κάποιες μικρές αλλαγές ε, όσον αφορά την κατηγορία στην οποία θα αλλάξουν ορισμένα κράτη-μέλη, γιατί διαπιστώνουμε ότι η εκτέλεση του προγράμματος είναι ικανοποιητική σε όλα τα κράτη-μέλη, επομένως οι τιμές που θα προτείνουμε στο προπολογισμό του 19 δεν θα αλλάξουν. Όσον αφορά τώρα τα μέτρα ε, Στήριξη της αγοράς. Δεν προβλέπουμε κατά τη διάρκεια του 2019 ιδιαίτερε δυσκολίες. Βεβαίως θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε εάν προκύψει κάτι το απρόπτο, χωρίς να φαίνεται κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Θα μείνουμε κάτω από το όριο και αυτό σημαίνει ότι θα δημιουργηθεί βεβαίως το αποθεματικό για την αντιμετώπιση των κρίσεων. Καταγράφουμε τις ε, επισημάνσεις που κάνετε σε αυτή την έκθεση, καθώς επίσης και τις επισημάνσεις που είχατε κάνει στο πλαίσιο της συζήτησης για το Omnibus και όταν θα, στις αρχές του Μαΐου η η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει την πρότασή της για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και αργότερα την πρότασή της, την η Επιτροπή για τη νέα ΚΑΠ. Θα δείτε πώς τις λάβαμε υπόψη μας και στην πράξη. Θα διατηρήσουμε επίσης κατά τη διάρκεια του 2019 να διατηρηθεί ένας υψηλός ρυθμός πληρωμών από τα διαρθρωτικά ταμεία, το 19, και θα πρέπει να ε, ακολουθήσουμε τι δεσμεύσει που έχουμε αναλάβει στο πλαίσιο προηγούμενων προγραμματισμών να κάνουμε πληρωμές προ τα κράτη-μέλη από τα ταμεία αυτά το 2019. Ε, Βεβαίω, όταν ε, θα είναι διαθέσιμα τα πιο συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία από τι διάφορε υπηρεσίε τη Γενική Διεθνή Αγροτική Ανάπτυξη. Όσον αφορά τώρα το σημείο 4 του προσχεδίου ψηφίσματό σα, όσον αφορά τα ειδικά μέτρα για την στήριξη των απορροκυπευτικών σε σχέση με το εμπάργκο. Δεν σκοπεύουμε να διατηρήσουμε αυτή την ιδιαίτερη στήριξη. Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από το ρωσικό εμπάργκο και ακούμε από τους εμπορευόμενους, από τους δραστηριοποιούμενους στον τομέα ότι έχουν βρει νέους τρόπους, άλλους τρόπους ε, εξαγωγής και οι εμπορευόμενοι για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που δημιούργησε το εμπάρκο. Βεβαίω υπάρχουν άλλα προγράμματα, όπω για παράδειγμα στο πλαίσιο του ΕΧΤΑ, που μπορούν να αξιοποιηθούν για διαρθρωτικέ αλλαγέ αν χρειαστεί. Όσον αφορά τώρα την επισήμανσή σα για τι επιπτώσει του Brexit, τι λαμβάνουμε υπόψη μα, όπω ορθά αναφέρθηκε, ο προπολογισμό του 2019 είναι Προπολογισμό ο οποίος έχει σχεδιαστεί για 28 κράτη-μέλη. Υπό αυτήν την βάση συζητούμε 28, συγγνώμη, κράτη-μέλη και τη Μεγάλη Βρετανία δηλαδή. Υπό αυτή τη βάση συζητούμε. Βεβαίω, εάν κάτι πολύ άσχημο συμβεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, γνωρίζετε ότι θα έχουμε όχι μόνο τη δυνατότητα, αλλά και την υποχρέωση να αποστείλουμε ε, πρόταση για διόρθωση του προπολογισμού, για τροποποίηση του προπολογισμού, ακόμα και κατά τη διάρκεια του 2019, αν χρειαστεί. Όσον αφορά το αποθεματικό για τις κρίσεις, στο σημείο 7 του ψηφίσματός σας προτείνονται κάποια επιπλέον μέτρα πολιτικής. Η ανακοίνωση μας για το μέλλον της Γεωργίας σας δίνει κάποιες ενδείξεις, όμως όπως σας είπα, ας αναμείνετε τις ανακοινώσεις της Επιτροπής το τέλη Μαΐου ε, για την ΚΑΠ και θα δείτε εκεί πιο συγκεκριμένα μέτρα για τους νέους αγρότες και άλλες, ε, άλλες τομείς που μας επισημαίνουν το σημαντικό στην πρότασή σας. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε κύριε Διευθυντά και ο λόγος και πάλι στον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συντάκτη της γνωματοτησής μας, τον κύριο Σίσο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ λακωνικά να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις προτάσεις τους και τους κοιόδης ηγητές και τους υπόλοιπους συναδέλφους που έλεγαν το λόγο. Και φαντάζομαι ότι με τις τροπολογίες θα εμπλουτίσουμε το κείμενο της γνωμοδότησης και θα απεικονίσουμε εύστοχα και γλαφυρά τις ανησυχίες της Επιτροπής Γεωργίας, που φυσικά είναι η προάσπιση των γεωργών και κτηνοτρόφων μας. Και θέλουμε για αυτούς να εξασφαλίσουμε έναν επαρκή προϋπολογισμό της κοινή γεωργικής πολιτικής για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Γεωργία να συνεχιστεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Βαλκάρ Σελσίσο. 27 Απριλίου λίγη προθεσμία για την υποβολή των απολογιών. Θα ψηφίσουμε στις 20 Ιουνίου γιατί η διορία για την υποβολή της γνωμοδότησης στην Αρμόδια Επιτροπή Προϋπολογισμών 21 Ιουνίου. Αυτά διεκπαιρεώσαμε την απογευματινή μας ημερήσια διάταξη. Είχαμε δυνατότητα για εκτενή συζήτηση που ήταν και απαραίτητη. γιατί αυτή η συζήτηση θα τροφοδοτήσει και τις εργασίες μας. Αύριο ξεκινούμε τη συνεδρία σε 9 με ψηφοφορίες, οπότε μην ξεχάσετε τις κάρτες ψηφοφορίας. Και το απόγευμα έχουμε κοινή συνεδρία με εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Το απόγευμα θα ξεκινήσουμε τη συνεδρία στις 2. Στις 2 παρακαλώ σημειώστε, σημειώστε το να μην το ξεχάσετε. Νωρίτερα από ό,τι συνήθως. 2 αύριο το απόγευμα και 9 το πρωί με τις ψηφοφορίες. Καλό σας βράδυ και ραντεβού αύριο στις 9 το πρωί. Χαίρετε.